Γεια σας και καλό απόγευμα. Είναι και μάτι πάλι η ημερήσια διαταξή, φορτωμένη. Καλά θα κάναμε λοιπόν να ξεκινήσαμε. ξεκινήσαμε. Να κοιτάξουμε λοιπόν το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι το 19. Διαχείριση τη διασυνοριακή κρίση στον τραπεζικό τομέα. Μία έκθεση και αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε επί του θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Uh, είναι πολύ δύσκολο το θέμα, αλλά νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει για να επιληθούν πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. It be Νομίζω, και δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω, ότι υπάρχουν θέματα που αποτελούν κινητήριο δύναμη του όλου θέματος. Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι τα συστήματα δεν είναι λειτουργικά και γι' αυτό χρειάστηκε να επιβιώσουμε με μεγάλη δυσκολία. Τα σχέδια αυτά ενέχουν πολύ υψηλό κόστος, ιδιαίτερα για τους φορολογούμενους και μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο παρενέβη για ποσό της τάξης των 850 δις στερλινών και θα κατανοήσουμε με το πέρασμα του χρόνου ποιο ήταν το άμεσο κόστος. Όμως, ακόμα και αν δεν έχουμε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία παρά μόνο ως ε, προβλέψεις, είναι δύσκολη η ποσοστοποίηση. Όπως ξέρετε, παρέλυσαν οι επιχειρήσεις, είχαμε αύξηση ανεργίας, ε, μείωση των εισοδημάτων λόγω υψηλής φορολόγησης και ούτω καθεξόποιος. και να είναι ο τελικός λογαριασμός βαραίνει ιδιαίτερα τους φορολογούμενους, υπήρξαν επιπτώσεις, βαριές επιπτώσεις στον τομέα απασχολησιμότητας και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να στραφώ σε μια δεύτερη σκέψη για πώς ε, μπορούμε να εξεύρουμε μια λύση. Δεν υπάρχει χρυσό χάπι για να χρυσώσει τα πράγματα. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα πακέτο το οποίο να είναι εξισορροπημένο. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε τους παλαιούς κανονισμούς. Έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες, προαπαιτήσεις κεφαλαίου για να καλύψουμε επιπρόσθετους κινδύνους, εισαγωγή ε, αναλογιών ρευστοποίησης και μηχανισμούς αναχώματος. Επίσης, θα πρέπει να καλύψουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εποπτείας, άρα η δική μου σχέση έχει μεγάλη σχέση με τις επόμενες εκθέσεις, τις εκθέσεις Μαργκάγιο, Γκίγκολτ, Σκίνερ και Γκουλάρ. Υπάρχει βεβαίως και μία άλλη επίπτωση που αφορά τη νέα αρχιτεκτονική του τραπεζικού συστήματος. Μιλάμε για επενδύσεις, τραπεζικές επενδύσεις και επενδύσεις λιανικής. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με αυτό το μεγάλο ανάχωμα νομοθεσίες, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μιας κρίσης. Εδώ όμως υπάρχει και το τέταρτο στοιχείο το οποίο υπησέρχεται δηλαδή η ευρωστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διασυνοριακή ε, διαχείριση της κρίσης. Και εδώ εμπλέκεται αυτό το έγγραφο. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα, δηλαδή όπως γνωρίζετε, όταν δούμε τι έχει επισυμβεί μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορισμένα ζητήματα μείζονο και θα πρέπει να προβούμε και σε μια αυτοκριτική. Βεβαίως χρειάστηκε παρέμβαση για να μην πέσουμε στον κρεμό, αλλά το σύστημα έτσι κι αλλιώ δεν ήταν αποδοτικό. Θα μπορούσαμε να, έχουμε, να τα έχουμε καταφέρει καλύτερα με χαμηλότερο κόστος για τους ε, φορολογούμενους. Υπήρχαν, υπήρξαν επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία. Τι έκαναν οι Ιρλανδοί, τι έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε στρεβλωμένο ανταγωνισμό και υπήρξαν και θέματα ως προς τα δικαιώματα των μετόχων. Από τη Northern Rock μέχρι πολλά άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είχαμε βεβαίως και νομοθετικές προκλήσεις, καθαρά νομοθετικές, και επήλθε μεγάλη σύγχυση και έλλειψη κατανόησης του νομικού πλαισίου των ε, εμπλεκομένων συμφερόντων και υπήρξε και πολύ ψηλός προστατευτισμός από πολλές κυβερνήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να μας επαναπασχολήσει το θέμα από πλευράς ε, ευρωπαϊκής πλαισίωσης. Μπορούμε να έχουμε μία ενοποιημένη ε, ενιαία αγορά σε σχέση με επιμερισμένα μέτρα των κυβερνήσεων. Εάν θέλουμε να προβούμε σε μια κοινοτική πλαισίωση, θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Μιλάμε για δεοντολογικής φύσης κινδύνους. Είναι ουσιώδες ζήτημα, βεβαίως και είναι, και θα πρέπει να μας απασχολήσει. Όμως, η κατάσταση που μας απασχόλησε θα ξανασυμβεί. Όλες οι κυβερνήσεις παρενέβησαν, διότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο κακό που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα να τονίσω ότι το θέμα δεν είναι να εγγυηθούμε την έλλειψη αποτυχίας. Θα, δεν θα πρέπει να προβούμε σε μία άσκηση ευθανασίας, αλλά αποκατάστασης. Θα πρέπει να διασώσουμε ό,τι μπορεί να διασωθεί έτσι ώστε να μην υπάρχει μία μετολίσθηση και σε άλλα στοιχεία του συστήματος. Αυτά τα τρία ζητήματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν, δηλαδή ο δεοντολογικός κίνδυνος πρωτίστως. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα της ενδεχόμενης ευθανασίας ή της επανόρθωσης και θα πρέπει να δούμε το θέμα επίλυσης θεμάτων αφαιρεγγιότητας έτσι ώστε να μην αναλάβει το συνολικό κόστος ο φορολογούμενος. Άρα τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι τα εξής. Υπάρχουν αναδυόμενες απόψεις και θα πρέπει να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ενιαία προσέγγιση εκκίνησης της παρέμβασης και να κατανοήσουμε σε ποιο επίπεδο θα επισυμβεί και θα πρέπει να βρούμε και τον κατάλληλο ρυθμιστή που θα παρέμβει. Επίσης, θα πρέπει να ορίσουμε ένα μίνιμουμ κανόνων που θα χρησιμοποιήσουμε σε μια πρωταρχική φάση αν θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο δύσκολες λύσεις. Θα πρέπει να συζητήσουμε ε, θέματα που αφορούν και την έκθεση Μαργκάγιο και θα πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό επιλύσεων με μια εποπτική αρχή και να απλουστεύσουμε κάπως τα πράγματα. Ένα λοιπόν ταμείο επίλυσης κινδύνων θα πρέπει να συσταθεί. Θα πρέπει όμως να συμφωνήσουμε σε μια σειρά κανόνων έτσι ώστε οι εποπτικές αρχές να μπορέσουν να επέμβουν, δηλαδή να υπάρχει ένα διευθυντήριο εποπτών. Ορισμένα ιδιαίτερα ζητήματα μας απασχόλησαν. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτό το πλαίσιο ορίζοντας την βαθμιαία σύγκληση των εθνικών νομοθεσιών με το διευρωπαϊκό. Ποια θα πρέπει να είναι η εμβέλεια της ρύθμισης. Θα πρέπει να έχουμε μία αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων και θα πρέπει να καλύψουμε και μη τραπεζικούς οργανισμούς που ε, επηρεάζουν την τύχη των τραπεζών αν έχουμε αυτό τον φορέα επίλυσης, θα μπορούσαμε να έχουμε και χρηματοδότηση αυτών των παρεμβάσεων και πώς ε, ορίζουν τα σχέδια καταθέσεων. Ποιες, ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί παρέμβασης. Πώς μπορούμε να εκινήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, αντικειμενικές αναλογίες που να μην ε, διακυβεύονται από τις τράπεζες που δημιούργησαν τους συστημικούς κινδύνους. Ποιους μηχανισμούς θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σε αυτές τις παρεμβάσεις. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα αρρωγής ρευστότητας ένα διατραπεζικό σύστημα γεφύρωσης. Θα πρέπει να έχουμε μία σειρά μηχανισμών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτούς τους, από αυτούς φορείς, τους παρεμβατικούς φορείς, αν θέλουμε να μπούμε στην ουσία της παρέμβασης. Μετά πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτές τις, ε, αυτά τα μέσα ή τους μηχανισμούς με βάση τα στοιχεία που σκιαγράφησε η Κομισιόν. Η Επιτροπή μιλά για έγκαιρη παρέμβαση, επίλυση και αφαιρεγγιότητα. Μπορούμε να έχουμε ήπια μέτρα, soft measures. Πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα της, ε, το θέμα της αφαιρεγγιότητας. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Σε αυτό το στάδιο των εργασιών θα ήθελα να υποβάλω αυτά τα ερωτήματα γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια σύγκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα σε αυτή την Επιτροπή αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ιστορική αυτή ευκαιρία έτσι ώστε να μειώσουμε ή να ε, ελέγξουμε τους ε, συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από την τραπεζική, την ανεξέλεγκτη τραπεζική αφαιρεγκιότητα. Και αυτό είναι το σημείο εκκίνησης. Θα ήθελα να ακούσω τον συνάδελφο, τον Μάικ Λίτζ, έτσι ώστε να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων και να γνωρίζω ποια είναι η άποψη της Επιτροπής, έτσι ώστε να υποβάλω την πρώτη το πρώτο προσχέδιο έκθεσης. Thank you um, Σας ευχαριστούμε πολύ, Ελίζα. Στην, ε, σε πρώτη φάση να ακούσουμε την κυρία Τέντα Χούμπνερα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, προέδρα και πρωτού περάσω στα συγκεκριμένα σχόλια για την πρόταση της κυρίας Φερέρα. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις γενικότερες, οι οποίες όμως είναι σημαντικές, θεωρώ, για τις, ε, νέα, τα νέα νομοθετήματα που συζητούμε σήμερα. Καταρχάς, ό,τι και να κάνουμε για τις χρηματοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη της οικονομίας μας. Και θα πρέπει πάντα να εξετάζουμε τον αντίκτυπο ενδεχόμενων νέων νομοθυμάτων στην ε, πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη ότι θα μπορούσε να είναι και αρνητικός ο αντίκτυπος. Δεύτερη παρατηρήση. Θεωρώ ότι οι χρηματοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που συζητάμε ε, καταδεικνύουν, αν θέλετε, μία μεσοπρόθεσμη βεβαιότητα σε ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο που θα επικρατήσει σε όλο τον κλάδο. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις μας αυτές δεν θα επηρεάσουν τον ανταγωνισμό με αρνητικό τρόπο και ότι φυσικά θα καταργηθεί ο ηθικός κίνδυνος. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Θεωρώ καταρχάς ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων για την αντιμετώπιση της κρίσης σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή του πλαισίου αυτού. Θεωρώ ότι θα πρέπει να καλύπτει και τον τραπεζικό κλάδο, αλλά και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ευρήματα. Επίσης, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει το ίδιο επίπεδο προστασίας για όλες τις οντότητες ε, και στη χώρα υποδοχής και στη χώρα προέλευσης. Να υπάρχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας. Όλα τα μέλη του ομίλου να την χάνουν τις ίδιες αντιμετώπισης. Επίσης, θεωρώ ότι είναι αδικαιολόγητο Να υπάρχουν τρεις, ότι πιστεύω ότι δικαιολογείται να υπάρχουν τρεις ε, φάσεις ε, και θεωρώ ότι είναι σημαντικά τα πλεονεκτήματα να υπάρχει, ε, του να υπάρχει ένα ε, σώμα ευρωπαϊκού επίπεδου που να προασπίσεται τα δικαιώματα όλων. Και φυσικά θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η ουδετερότητά του και η ανεξαρτησία του. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Εξυγίανσης. Το βασικό θέμα, όπως είπε και η Ελίζα, είναι από πού θα χρηματοδοτηθούν οι δαπάνε. Αν οι χρηματοδοτηθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή οι μικρές τράπεζες θα δυσκολευτούν. Επίσης αναφέρεται η δυνατότητα σύνδεσης με τα σχέδια εγγύησης καταθέσεων. Αν ε, επιλέξουμε τη λύση των κυβερνήσεων, δεν θα πρέπει να εξετάσουμε μόνο τη δυνατότητα εκδοτήσεων, αλλά και των κρατικών δανείων. Τελευταίο σχόλιο. Το ανέφερε λίγο και η Ελίζα. Είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την συνοχή σε ό,τι αφορά το πλαίσιο αυτό της κρίσης και όλων των ε, κανόνων που συζητιούνται και που εισάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά να ληφθούν υπόψη και οι αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ να ακούσουμε και τους υπόλοιπους κοιόδης. Η κυρία Σφίμπορτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να συγχαρώ την Ελίζα για τη δουλειά που έκανε και για την προσέγγιση της σε ένα πολύ πολύπλοκο θέμα. Καλωσορίζω πραγματικά το γεγονός ότι διοργάνωσε με συζητήσεις στο Στρασβούργο ήδη πριν από κάποιες εβδομάδες με τους κοιόδης. Είναι πολλά και ιδιαίτερα περίπλοκα τα θέματα και θεωρώ ότι ιδιαίτερα σημαντική είναι η ιδέα της εναρμόνισης των νόμων περί φρεγιότητας ε, στην Ευρώπη. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το δυνατότητα ε, χορήγησης ε, εξαιρέσεων. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες να εξετάσουμε. Καλωσορίζω την ε, πρόταση που αφορά το σώμα των εποπτών. Είναι σημαντικό γιατί πολλές τράπεζες έχουν έδρα σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχουν δραστηριότητες και στην Ασία ή στην Αμερική. Επίσης έχουμε πολλές τράπεζες σε μέτρα την Αμερική που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το σώμα των εποπτών θα λειτουργεί σωστά. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε κάτι αντίστοιχο του άρθρου 11 ε, του Αμερικανικού νόμου σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις αυτές. Είναι σημαντικό, ωστόσο, οι μέτοχοι να γνωρίζουν ότι οι επενδύσεις τους διατρέχουν κίνδυνο σε οποιαδήποτε μορφή. Και νομίζω ότι αυτό που κατέστησε σαφές στην έκθεση αυτή είναι η ανάγκη να εξετάσουμε τους κινδύνους. Θα πρέπει να καταργήσουμε αυτή την οτροπία ότι κάποιο ίδρυμα είναι υπερβολικά μεγάλο και δεν μπορεί έτσι να πτωχεύσει. Θα πρέπει αυτό πραγματικά να εκλείψει. Και θα ήθελα να καλέσω τα μέλη της Επιτροπής μας να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δώσουν μια να θέσουν μια εξωτερική μελότη σε ό,τι αφορά ε, τέτοιες επενδύσεις για να ξέρουμε τι μέγεθος θα μπορούσε να αποκτήσει μια τέτοια ευρωπαϊκή θεσμική τράπεζα. Θα μπορούσαμε να σώσουμε μια ολόκληρη τέτοια τράπεζα όπως η Deutsche Bank για παράδειγμα ή ένα τμήμα αυτής που αυτό θα συνεπαγόταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει απόθεμα δισεκατομμυρίων ευρώ. Και σε τι α, επενδύσεις θα έπρεπε να προβεί μια τέτοια τράπεζα και θα ήθελα να εξασφαλίσω ότι η Επιτροπή μας θα καταρτήσει μία έκθεση που θα είναι ρεαλιστική σε ό,τι αφορά με που αφορά τέτοιες πανευρωπαϊκές επενδύσεις. Μιλήσαμε για τις εγγύησεις καταθέσεων. Θα πρέπει να σας πω ότι έχω κάποιες αμφιβολίες. Θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να προστατεύουν τους καταθέτες. Δεν θα πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση να διατρέχουν κίνδυνο αυτά τα στοιχεία. Γιατί οι καταθέτες τελικά αυτοί που θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο σε τέτοιες ε, περιπτώσεις κρίσης. Συνοψίζοντας λοιπόν, θεωρώ ότι το σέμα των εποπτών θα πρέπει να συμμετάσχει και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις Αμερικανικές τράπεζες. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μια έκθεση ε, εφικτότητας για τα ταμεία αυτά και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε τέτοιες εγγύσεις καταθέσεων με οποιοδήποτε επενδυτικό ταμείο εξυγίανσης για να μην ε, διακυβεύονται αυτά τα κεφάλαια. Ο κύριος Όλη Σμιτ. Ε, Ευχαριστώ. Να συγχαρώ και εγώ την Ελίζα Φερέιρα για το εγγραφό τη. Ε, φυσικά, όπως πάντα, κάνει ενδιαφέρουσες προτάσεις. Ε, όχι πάντα, σχεδόν πάντα. Πάντως είναι ειλικρινής και ακόμη και από ένα φιλελεύθερο κάποιος θα μπορούσε, από πλευράς φιλελευθέρων θα μπορούσαμε να τις ενστερνιστούμε τις ιδέες της κυρίας Φερέιρα. Νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε συνένεση ούτως ή άλλως και να αντλήσουμε και πολλά διδάγματα από αυτά που έχουν συμβεί. Ε, στην Επιτροπή μας ε, βλέπω μια υπερβολική προθυμία να γίνονται προτάσεις, να θεσπίζονται νέα νομοθετήματα και καμιά φορά θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι δεν χρειάζονται απαραίτητα κανονισμοί όταν τους βλέπουμε ως αυτό σκοπό καλύτερους κανονισμούς ε, χρειαζόμαστε, ποιοτικότερους ε, κανονισμούς Το πρωί συζητούσαμε 1.700 τροπολογίες Μα 1.700 τροπολογίες δίνουν την εντύπωση ότι θα εκπονήσουμε καλύτερη νομοθεσία, έναν αποτελεσματικότερο κανονισμό. Πολύ αμφιβάλλω. Εξαλλού χρειάζεται συνένεση, όπως σας έλεγα, όλων των ε, πολιτικών ομάδων ε, και να συγκεραστούν 27 διαφορετικές παραδόσεις. Αφήστε ότι υπάρχουν και πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς εκτός των 27 της Ένωσης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην ε, θεσπίσουμε ένα πλαίσιο που τελικά θα αποβεί επιζήμιο για την αγορά η οποία αγορά ψάχνει το φως στην άκρη της σύραγγας. Πολιτικός πόσο δεν είναι σοφό αυτό που θα πω, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον ε, κάποιοι να το σκεφτούν. Τελικά πρέπει να αποκτήσουμε ένα μέτρο για να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των προτάσεων της Επιτροπής μας. Σχετικά με τον οργανισμό εξυγίανσης και αυτό το ταμείο εξυγίανσης, ε, νομίζω ότι μπορεί να παίξει κέριο ρόλο. Όπως ακούσαμε, είναι σημαντικό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην δημιουργήσουμε ένα τέρας, ένα Φρακενστάιν. Αυτά τα τεράστια ταμεία χρειάζονται και παρακολούθηση. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι προτείνουμε. Εγώ προέρχομαι από μικρή χώρα που αντιμετώπισε τέτοια πελώρια προβλήματα δεκαετία του 90 και ήμουν στην μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών και τότε είχαμε 500% επιτόκια και είχε αυξηθεί μέχρι 2.000% και καταφέραμε τελικά να λύσουμε την κρίση. Και η κυβέρνηση την οποία στηρίζω τώρα τουλάχιστον έχει ένα ε, σχέδιο σταθερότητας για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ένα ταμείο σταθερότητας. Ο Σουηδός Υπουργός Οικονομικών Έλαβε πρόσκληση από τον πρόεδρο Ομπάμα. Δεν ξέρω αν καθησυχάζει αυτό κάποιο εδώ στην Επιτροπή μα, Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, ε, ε, οι ιδέε που έχει η Σουηδία θεωρούνται καλές τη είπα. Το θέμα είναι να φτάσουμε το 2,5% του ΑΕΠ σε κάποια χρόνια και θα χρησιμοποιήσουμε τις αμοιβέ από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από τράπεζες. Επίσης υπάρχουν κονδύλια από τον εθνικό προϋπολογισμό, αλλά ο στόχος είναι ίδια, ο ίδιος ο κλάδος να ε, χρηματοδοτήσει. Όλοι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που καλύπτονται από την εθνική ε, σχετική νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχει τέλος ε, σταθερότητας που χρηματοδοτεί το Ταμείο. 0,036% το χρόνο. Αυτό είναι το τέλος και εισπράτεται από, κάποιες, από, από κάποια από τα στοιχεία του παθητικού των χρηματοπιστωτικών φορέων και χρησιμοποιούνται όλα εκτός από τις ομολογίες ό,τι συμπεριλαμβάνεται στην κεφαλαιοχική βάση για τον υπολογισμό του τέλους και οτιδήποτε δεν έχει σχέση με συναλλαγές που σχετίζονται με δάνεια. Και υπάρχει και ένα, ένα συνδυασμό με το σύστημα των εγγυήσεων για τις καταθέσεις. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτή την ιδέα στα πλαίσια του αξιο... της ε, αξιολόγησης αντικτύπου. Γιατί υπάρχει και το ζήτημα του καταμερισμού των βαρών. Το να αφήσουμε τις τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς να χρηματοδοτήσουν το σύστημα είναι καλή ιδέα κατά τη γνώμη μου. Ε, δηλαδή η ανοικοδόμηση των τραπεζών ε, ε, και όχι οι φορολογούμενοι θα συμβάλλουν στο σύστημα. Πανευρωπαϊκή τώρα χρηματοδότηση. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει αυτό τώρα να συνιστά προτεραιότητα γιατί δύσκολα θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε αυτό το θέμα με τα εθνικά συστήματα εποπτείας αλλά θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο και να έχουμε κάποια πρόταση, τουλάχιστον ένα πλαίσιο Το χρειαζόμαστε κατά τη γνώμη μου. Ελίζα, ε, εν κατακλείδη θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό το έγγραφο που εκπώνησες και τα επιμέρους σημεία που τονίζεις είναι ενδιαφέροντα και θα πρέπει να τα εξετάσουμε περαιτέρω. Πάντως επαρκεί η πρότασή σου δεδομένου του πλαισίου των συζητήσεών μας και ακόμη και εγώ που είμαι φιλελεύθερος σε αυτό το συγκεκριμένο στάδιο αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζονται κανονισμοί στην αγορά. Εντάξει τώρα το είπα αλλά μην υπερβάλλετε. γιατί δεν πρέπει να σκοτώσουμε την αναδυόμενη αγορά. Ευχαριστώ όλοι, ο όταν ε, επανήλθα χτες, σκέφτηκα. Α, άλλαξε προς το χειρότερο το πνεύμα της Επιτροπής. Χάρη στον όλη τώρα ε, έχω λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη. Ας ε, συνεχίσετε για να μην αναθεωρήσω. Χτες άκουσα τα ίδια από αυτά που ξέρω από την εμπειρία μου και έχω κάποιες αμφιβολίες, αλλά ε, πάντως... Rethinking uh, Ας ε, ξανασκεφτούμε τι σημαίνει ο πραγματικός, ε, τι πρέπει να σημαίνει ο πραγματικός φιλελευθερισμός και ο πραγματικός συντηρητισμός. Ευχαριστούμε για αυτή την αναβίωση και ξαναλέω ότι έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο μέλλον με αυτά που άκουσα τώρα. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για αυτό το έγγραφο. Είναι πραγματικά καλή βάση για τις συζητήσεις. Ε, συμπεριλαμβάνονται όλα τα βασικά σημεία μπορούμε να συνεργαστούμε ε, σε αυτή τη βάση και θα κάνω μόνο δύο παρατηρήσεις. very Πρέπει να αναφέρουμε Ρίτα, ότι ο τραπεζικός τομέας έχει δημιουργήσει οικονομικό κόστος στο εξωτερικό. Τι εννοώ. Δηλαδή δεν έχουν συνυπολογιστεί στο σύστημα καθορισμού τιμών αυτά τα νέα, αυτό το νέο κόστος δεν έχει συνυπολογιστεί στον καθορισμό των τιμών του ίδιου του συστήματος. Είναι εξωγενές κόστος. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει αυτό. Πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος ε, στη διαμόρφωση των τιμών για να επανορθωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται αυτό τόσο ώστε να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις ε, μιας φιλελεύθερης οικονομίας. Νομίζω ότι ευσταθεί αυτό το επιχείρημα. Κυρίως όταν συζητούμε για το Ταμείο Εξυγίανσης. Σχετικά με τη σύσταση του Ταμείου, θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις στην έκθεση για την Τραπεζική Αρχή και για την ΕΣΜΑ. Οπότε δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Ε, θα σχολιάσω αυτά τα θέματα όταν φτάσουμε σε αυτό το θέμα. Ιστορικά έχουμε διασώσει μεγάλες τράπεζες Θυμηθείτε τι έγινε με τα κεφάλαια διστάθμισης κινδύνου τη δεκαετία των 90 στη ΣΥΠΑ. Υπήρχε ανάγκη διάσωσης. Τώρα τι άλλο μπορεί να γίνει. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν ε, θα ε, υπάρξει διάσωση, σχέδιο διάσωσης ε, για τις τράπεζες. Όπως είπατε εσείς, αλλά μας δείχνει η ιστορία ότι αν δεν υπάρξει σχέδιο διάσωσης θα, θα προκύψει ακόμη υψηλότερο εξωτερικό κόστος, εξωγενές κόστος. Ποιο είναι το δίδαγμα. Ναι, μεν να συστήσουμε το ταμείο, αλλά να μην υπάρχει κανόνα σχετικά με το πότε θα χρησιμοποιηθεί ε, το Ταμείο για ψυχολογικούς λόγους. Έτσι. Ε, οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν, πρέπει να, ε, φορείς δεν πρέπει να ξέρουν πότε θα χρησιμοποιηθεί αυτό το Ταμείο. Και υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ αυτής ε, της ε, στάσης ότι ακόμη και αν υπάρχει το ταμείο πρώτα πρέπει να πληρώσουν οι ιδιοκτήτε τη Τράπεζα και μετά ε, να αναλάβουν άλλοι το κόστος αλλιώς από πλευράς φιλελεύθερης ορθοδοξίας δεν μπορεί να ευσταθεί προσπάθεια που κάνουμε. Ευχαριστούμε η Δίκη. Ναι, συγγνώμη, η Βίκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ξεκινώ από την αρχή ότι θεωρώ ότι τα ιδρύματα θα πρέπει να έχουν ε, την δυνατότητα, αν θέλετε, να αποτυγχάνουν, γιατί αν δεν αποτύχαναν θα σήμαινε αυτό ότι είχαν υπερβολική στήριξη. Άρα χαίρομαι που αυτό αποτελεί το σημείο κίνησης, ο ηθικός κίνδυνος. Δεύτερο σημαντικό θέμα είναι το όλο θέμα των διασυνοριακών πτωχεύσεων και των νομικών αγωγών. Και επειδή ε, εγώ συμμετείχα σε τέτοιες προσπάθειες αποτροπής ε, πτώχευσης, ξέρω τι σημαίνει ε, να υπάρχουν τέτοιες ε, περιπτώσεις. Και έχοντας ε, δει πόσο δύσκολο είναι να καταλήξουμε σε γενικότερη συμφωνία για τα λογιστικά πρότυπα ουσιαστικά, ε, πραγματικά ε, θεωρώ ότι είναι τεράστια πρόκληση να υπάρξει γενικά συμφωνία για τα πρότυπα πτώχευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπαμε και το πρωί, δεν μπορεί να είναι το φυλακή ούτε ο χειρό θα πρέπει να σκεφτούμε παγκόσμια, όχι μόνο στο στενά πλαίσιο της Ευρώπης, αλλά θα ήθελα να εξετάσουμε και κάποιες άλλες διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν πρωτού περάσουμε σε πτώχευση, πρωτού χρειαστεί εξυγίανση. Να, όσο είμαστε στη φάση της ανάκαμψης και στην φάση της ανάκαμψης θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχει θέληση διατήρησης της ε, τράπεζης. Και κάποια εντρήματα θα πρέπει να έχουν εξετάσει τα μέτρα κατεπίγουσας ανάγκης προτού περάσουν στην φάση της τελικής και ολοκληρωτικής πανολευθρίας. Και θα πρέπει να ε, ξεκινήσουν τη διαδικασία ανάκαμψης τους προτού περάσουν απαραίτητα στη φάση εξυγίανσης. Ανησυχώ κάπως για το αν χρειάζεται ε, ένας επιπρόσθετος οργανισμός. η ποτέ χρειάζεται ένας οργανισμός εξυγίανσης. Εγώ θα θεωρούσα ότι καλύτερα να κατανεμηθούν αυτές οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες σε ήδη υφιστάμενα συστήματα και ιδρύματα. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο στη τελική ανάλυση θα λειτουργεί. Η άλλη συζήτηση που θα πρέπει να έχει γίνει πριν ε, από την πτώχευση είναι το θέμα του δεσμευτικού κεφαλαίου. Θα πρέπει δηλαδή κάποιο από το χρέος να έχει μεταφερθεί σε equities. Ακόμα και αν πρόκειται για φορολογούμενους ή για ιδιωτικέ εταιρείε που θέλουν equities, θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία για την εξυγίανση του ισολογισμού. Και εδώ θα βοηθούσε το δεσμευτικό κεφάλαιο. Και σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Ευχαριστώ, κύριος Σκίνερ, Πείτε, Σκίνερ. Η Ελίζα μας συνέταξε ένα προκλητικό έγγραφο, το οποίο είναι εξαιρετικό, έχει εξαιρετικά στοιχεία. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Καταρχήν, Ελίζα, προβλέπεις ή ξέρεις κατά πώς θα υπάρξει, θα ανακύψει τομεακή νομοθεσία και πώς θα εισαχθεί. Γιατί αυτό σε απασχόλησε διαχρονικά, το συζήτησες και με άλλους, τι χρονοδιάγραμμα προβλέπεις για την εισαγωγή μιας ειδική νομοθεσίας. Μπορεί να γίνει νωρίτερα παρά αργότερα, γιατί υπάρχουν πολλές πιέσεις επί του παρόντος. Ο Ζαν Πολ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ ε, Λίζα και να την ε, ευχαριστήσω θερμά διότι πρόκειται για μία ε, δύσκολη αποστολή, να μην πω ακατόρθωτη αποστολή. Εγώ θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις ληστικής φύσης σε ένα τέτοιο θέμα τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να συνταχθεί μία έκθεση, μία μελέτη, κάτι το οποίο δεν μου αρέσει ιδιαίτερα ή θα πρέπει να διευρύνουμε τη συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να είμαστε γρήγοροι ότι θα γίνει λόγος είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Ίσως θα πρέπει να πούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες για να δούμε τι μπορεί να γίνει με τέτοια ε, ταμεία εγκυοδοσίας και νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να ανταποκριθούμε με τα μέσα που έχουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι μία ευρωπαϊκή ρύθμιση και μία ευρωπαϊκή εποπτική αρχή. Συμφωνώ με την κυρία Φόρτ που λέει μην χρησιμοποιήσουμε, μην δημιουργήσουμε άλλον ένα φορέα. Εάν έχουμε μία αρχιτεκτονική εποπτείας που να έχει τα κατάλληλα μέσα και τις αρμοδιότητες, τότε θα έχουμε φτάσει σε μία επίλυση. Τα εθνικά, τα κράτη-μέλη δεν δέχονται πάντα μία ευρωπαϊκή εποπτική αρχή. Αντιστέκονται αλλά δεν αποφασίζουν μόνοι τους ε, οι Υπουργοί. Έχουμε και εμείς το δικό μας λόγο. Σήμερα καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες ε, υπό αυτή την οπτική γωνία και θα πρέπει να καταβάλουμε και εμείς προσπάθειες μέσα στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής που να είναι αποτελεσματική, πραγματιστική και η οποία θα μας προσδώσει τα μέσα να ανταποκριθούμε στην κατάσταση, διότι οι εποπτικές αρχές είναι πλέον αρμόδιες. Υπάρχει και η τεχνική πλευρά του θέματος. Ας τους δώσουμε τις αρμοδιότητες λοιπόν, γιατί διαφορετικά ε, αν δεν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε σε επίπεδο 27 θα το καταφέρουμε παγκόσμιο. Ο Γκαρθία το ανέφερε αυτό στις εκθέσεις του. σε σχέση με τον συστημικό κίνδυνο και της, ε, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες και έτσι, έτσι ώστε η Ελίζα να μπορέσει να κάνει μια συγκεφαλαίωση όλων αυτών των τάσεων και να μας πει ότι το πρότεινε και τελικά υλοποιήθηκε, πραγματώθηκε η Σίλβι Γκουλάρ και εγώ θα θέλαμε να πάρουμε και ο Γκαρθία Μαργκάγιο νομίζω θέλει το λόγο. Κλείνω τον κατάλογο, αλλιώς δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Χούμπνε ότι υπάρχουν μακροοικονομικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα ως προς τις ε, προαπαιτήσεις κεφαλαίου. Και αυτό που έχει σημασία είναι ε, να δούμε τι κεφαλαϊκές απαιτήσει υπάρχουν ή κεφαλαϊκές προαπαιτήσει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε άλλες πλαισιώσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πριν ε, προβούμε σε μία διάσωση. Η μεταφορά στοιχείων ενεργητικού διασυνοριακά θα πρέπει να είναι ένα από αυτά τα μέσα. Ίσως είναι δύσκολο και ίσως είναι πολύ πιο δύσκολο όταν φτάσουμε στο στάδιο της πτώχευσης αλλά υπάρχουν πολλές ιδέες για να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μια διασυνοριακή προσέγγιση και όχι μόνο να κινούμαστε σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι στην έκθεσή σου μίλησες για την κάλυψη όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά βεβαίως θα είναι πολύ δύσκολο. Μίλησες για το phasing, το οποίο είναι κρίσιμης ε, σημασίας αν θέλεις να συμπεριλάβεις τις ασφαλιστικές εταιρείες, η κατάσταση είναι διαφορετική. Γιατί δεν ξέρουμε τι αξιώσεις θα προβληθούν. Άρα το χρονοδιάγραμμα είναι διαφορετικό. Άρα η διάσωση ίσως να μην είναι, μια συγκεκριμένη μορφή διάσωση ίσως να μην είναι η σωστή. Προσπαθούμε να έχουμε ιδέες για μια αξιολόγηση, ιεράρχηση ε, μέτρων για μια κατάσταση πριν από την πτώχευση, για μια ε, κατάσταση προπτωχευτική και ιδιαίτερα να δούμε τι αξιώσεις προβάλλονται. Διασυνοριακά θα δούμε ποιοι κατέχουν ε, ε, ασφαλιστικά συμβόλαια και όταν μιλάμε για policy holder δεν εννοούμε, ε, δεν μιλάμε μόνο για κατάσταση καθαρά εθνική και αυτό το είδαμε με την ασφαλιστική εταιρεία Equitable Life. Και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό καθεστώς για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή μόνο για τράπεζες και μετά να κινηθούμε σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Υπάρχει όμως ε, μία σύγχυση ως προς την εξηγίαση ε, εταιριών, corporate resolutions. Και εάν δούμε αυτές τις ε, πτυχές εν συνόλο, τότε θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μια κατάσταση κρίσης, διότι ε, πολλές φορές δεν μπορούμε να διασώσουμε τα πιστοτικά ιδρύματα σε μια προπτωχευτική φάση. Δεν ξέρω πώς, ε, ε, μάλλον τι κατανομή θα μπορέσει να υπάρξει, κατανομή ευθυνών ή μέτρων αλλά η Επιτροπή θα μας προτείνει και άλλα μέτρα, ιδιαίτερα σε σχέση με ένα τέλος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ίσως προβλέψουμε και άλλα μέτρα. Στο μεταξύ, η Σιλβία έχει το λόγο στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ελίζα για αυτή την εργασία η οποία είναι πολύ σημαντική. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε τη διασυνοριακή κατάσταση διότι όταν συζητάμε με ορισμένου φορείς έχουμε την εντύπωση ότι η διασυνοριακή ε, φάση έχει συρρυκνωθεί και νομίζω ότι μέσα στο πακέτο της εποπτείας αυτό είναι ένα ε, στοιχείο μίζωνο σημασίας δηλαδή εποπτεύουμε και δεν ξεχνάμε τον ενιαίο χαρακτήρα της αγοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για να απαντήσω στον Ζαν Πολ, δεν πρέπει να προτρέχουμε και να το αναθέσουμε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο το όλο θέμα. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουν τα εμπλεκόμενα κράτη. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι κάνουμε εμείς. Αυτό είναι, αποτελεί μία από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και αν θέλουμε και εμείς να έχουμε ειδικό βάρος, δεν θα πρέπει να δεχτούμε έξωθεν επιβαλόμενες λύσεις. Θα πρέπει να έχουμε μία συνεκτική προσέγγιση και η Ελίζα Φερέιρα μας δίνει ορισμένες απαντήσεις και αυτό αφορά και την έκθεση ε, Μαργκάγιο και Γκίγκολτ. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Ελίζα γιατί έχουμε μια συνεκτική, μας έδωσε μια συνεκτική προσέγγιση που είναι ιδιαίτερα ε, χρήσιμη. Μαργκάγιο. Ε, τέσσερα σημεία θα ήθελα να θίξω και θα τα θίξω όταν μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών στη συνέχεια, ως προς τη δική μου έκθεση δηλαδή. Νομίζω ότι η έκθεση Φερέιρα είναι πολύ χρήσιμη Ε, θα ήθελα να πω προς τον συνάδελφο Σβεν ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να φτάσουμε σε αίσιο πέρας. Θα πρέπει δηλαδή ε, να λάβουμε υπόψη τον πολιτικό λόγο τον οποίο προτάσουμε. Υπάρχουν ε, δύο μορφές προσέγγισης καταρχήν να δούμε τι θα κάνει το Συμβούλιο έτσι ώστε να προτρέξουμε και να προβάλλουμε μια γρήγορη διαπραγμάτευση και η δεύτερη προσέγγιση είναι να δούμε τι σημαίνει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς μπορούμε να παρέμβουμε. Ε, εμείς προβάλλουμε την θέση μιας ευρωπαϊκής οικοδόμησης και εδώ ξέρουμε ότι θα έχουμε την αντίσταση των εταιριών που δεν θέλουν να αλλάξει το status quo. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και υπάρχει και η αντίσταση των κυβερνήσεων, οι οποίες δεν θέλουν να εκχωρήσουν αρμοδιότητες. Ε, υπάρχουν, υπάρχει αυτό το διτό δέλεαρ δηλαδή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και όπως είπε και ο συνάδελφος «impossible c'est pas français». Δηλαδή οι Γάλλοι δεν πιστεύουν στο ανδύνατο του οποιοδήποτε εγχειρήματο. Η Ελίζα γνωρίζει ότι πάντα θα είμαι στη διάθεσή της για να φτάσουμε σε μία συμφωνία. Συμφωνία που θα πρέπει, για την οποία θα πρέπει να προτρέξουμε. Θα πρέπει να δούμε το διαχειριστικό πλαίσιο της ε, κρίσης. Χτες της ε, Financial Times είδα τι ε, ακριβώς προβλέπουν ορισμένοι ε, αναλυτές όπως ο Σόρος που λένε ότι θα πρέπει να προτρέξουμε ορισμένων συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να ληφθούν. Να προτρέξουμε έτσι ώστε να προβάλλουμε κάτι άλλο, ένα αντίπαλο δέος. Και αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε είναι να πούμε ότι εμείς θα ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας όπως ακριβώς ορίζονται. Η Ελίζα θα ήθελα να επανέλθει και να ανακεφαλαίωσει για δύο λεπτά, όχι πιο πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από αυτές τις εξαιρετικά πλούσιες παρεμβάσεις δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Θα τονίσω μόνο ότι μπορώ νομίζω να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πολιτική βούληση στο κοινοβούλιο μας για να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα παρά τις δυσκολίες και ότι δημιουργείται ένα πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα μας εδώ στην ε, Επιτροπή μας παρά το ότι υπάρχουν διαστάσεις απόψεων ε, λόγω πολιτικής κατεύθυνσης. Ε, πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για να συνεργαστούμε στο γη όσο καλύτερα μπορούμε. Και δεν θα είναι αυτό σκοπό η νέα νομοθεσία. Μόνο αν χρειάζεται θα την θεσπίσουμε και θέλουμε και αναλογικά μέτρα για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Πρέπει να είμαστε λογικοί και να αξιολογήσουμε την ικανότητα υλοποίησης αποτελεσματικών μέτρων που ε, λυσιτελών μέτρων να μην αναλαμβάνουμε υπερβολική δράση, να χρησιμοποιήσουμε τις ευθερίες που έχουμε και να κάνουμε μόνο ό,τι χρειάζεται. Κάτι άλλο τώρα με το οποίο θα κλείσω είναι ζωτική σημασία να έχουμε ε, ένα συνεκτικό προϊόν με όλες αυτές τις επιμέρους νομοθετικές πράξεις που εξετάζουμε. Αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό που πρέπει να κάνω εγώ τώρα μου φαίνεται να συνεχίσω το διάλογο με τους συναδέλφους που ακούσαμε και με τους υπολείπους, από τον κλάδο μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πανεπιστήμια, τους ερευνητές. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, τη θέσπιση μιας ε, συνεκτικής νομοθετικής πράξης. Έχουμε έναν απότερο στόχο, σταδιακά θα φτάσουμε εκεί. Με λογικό τρόπο, αλλά με αποφασιστικότητα. Η τέχνη της ισορροπίας. Αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε, αλλά από αυτά που άκουσα ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάντως ε, όλους όσους παρενέβησαν για τη διαθεσιμότητά τους σιγά σιγά Νομίζω θα καταλήξουμε σε μια λογική και αποτελεσματική πρόταση. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να δαπανίσω άλλο χρόνο, Πρόεδρε. Τα αυτά και μένω. Και διαδικαστικό. Ζητάμε να εκπονηθεί η έκθεση γιατί μιλάμε για 2,5% του ΑΕΠ βάσει της Σουηδικής πρότασης για 15 χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα 350 δις ευρώ για φέτος. Ε, νομίζω θα βοηθήσει μια αξιολόγηση αντικτύπου, Πρόεδρος. Ξέρετε, οι συντονιστέ θα αποφασίζουν αυτά, θα, θα, θα συζητηθεί το θέμα, αλλά μπορούμε να εργαστούμε προπαρασκευαστικά για να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Το χρονοδιάγραμμά μας για αυτή την έκθεση είναι 12 Απριλίου για την εξέταση του σχεδίου έκθεσης, καταληκτική για τις τροπολογίες 31 Απριλίου, εξέταση ε, τροπολογιών 1 Ιουνίου, 22 Ιουνίου ψηφοφορία στην Επιτροπή και πρώτη ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το ε, προτινόμενο χρονοδιάγραμμα. Περνάμε τώρα στο σημείο 4. Πρώην σημείο 4 για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Εμμανουέλ Γκαρθία Μαγκάλο και πάλι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Έχουν διατυπωθεί, έχουν ανακύψει 16 τροπολογίες και δέχομαι 12 από αυτές και έχω πρόβλημα με τέσσερις και θα σχολιάσω μόνο αυτές τις τέσσερις. Δεν ε, έχει νόημα να σας πω γιατί δέχομαι τις υπόλοιπες δώδεκα. Δηλαδή τις δέχομαι γιατί μου φαίνονται πολύ καλές και αυτό αρκεί. Σε σχέση με αυτές εκείνες που δεν δέχομαι, θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια έτσι ώστε να αντιδράσουν και οι υποβάλλοντες. Η πρώτη που δεν δέχομαι είναι η τροπολογή 28 Εστρέζεκ που αναφέρεται στο άρθρο 22.1. Προτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με, την, με το καλό ε, διαχειριστικό πλαίσιο του ΦΠΑ και η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να είναι αυτόματη. Δηλαδή μία αυτόματη διαδικασία αλλά προγενέστερη έγκριση από τα κράτη-μέλη. Πιστεύω όμως ότι σε αυτή την περίπτωση ε, θα έπρεπε να διαχειριστούμε τον ΦΠΑ κατά επιμερισμένο τρόπο γιατί αυτό έχουμε εισαγάγει στο πρώτο μέρος της τροπολογίας για να συρρυκνώσουμε κάπως αυτόν τον αυτοματισμό. Νομίζω ότι πρόκειται για μία ρήτρα διασφάλισης που είναι επαρκής. Άρα, αν ένα κράτος μέλος δεν γνωρίζει ότι γίνεται ε, μία παρέμβαση που του περιορίζει εξουσίες, αυτό δεν θα ήταν καθόλου καλό. Η δεύτερη τροπολογία που δεν δέχομαι είναι η 31 που αναφέρεται στο άρθρο 35. Αυτή η τροπολογία προτείνει την διοικητική και λειτουργική αρρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στα πλαίσια του ΕΡΟΦΗΣ για να βελτιώσουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τεχνική υποστήριξη για πολλά άλλα ζητήματα, τα οποία ορίζονται στην ε, πρόταση η οποία μας απασχολεί. Η επόμενη που δεν δέχομαι είναι η 32 που αναφέρεται στο άρθρο 35. Δηλαδή που είναι το ακριβώς αυτό που είπα πριν. Δεν δέχομαι η αρχή υποβολής της πρότασης του συντονισμού να είναι η Επιτροπή. Γιατί μπαίνουμε σε μία διαδικασία καθαρά διακυβερνητική, όπου μιλάμε για προβλήματα τα οποία αναγνωρίζουν και με τα οποία ταυτίζονται τα, κράτα, τα κράτη-μέλη. Άρα το ΕΡΟΦΙΣ θα πρέπει να μπορεί να παρέμβει έτσι ώστε να μην υπάρχει απάτη ή να εξαλειφθεί η απάτη ως προς το ΦΠΑ. Η τελευταία τροπολογία αναφέρεται στον ε, καλό φίλο Όλε Σμιτ είναι η 36. Δεν τη ούτε εκείνη. Ο κύριος ε, Σμιτ μας λέει ότι εάν χρειαστεί η Κομισιόν θα ε, προβεί σε επιμελητιακή βοήθεια στα κράτη-μέλη. Εδώ θα πρέπει να δούμε ποιος θα ορίσει αυτή την πλαισίωση. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Γι' αυτό θα προτιμούσα την διατύπωση της Κομισιόν που λέει ότι η Κομισιόν μπορεί να διαθέσει στα κράτη-μέλη μέσα και ούτω καθεξής, όταν το κρίνουν σκόπιμο τα κράτη-μέλη ή η Επιτροπή. Και εδώ μιλάμε για την καταπολέμηση της απάτης αποκλειστικά. Αυτές είναι οι τέσσερις τροπολογίες που δεν μπορώ να δεχτώ. Όλες τις υπόλοιπες ε, μπορώ να τις δεχτώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο, ο οποίος με βοήθησε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε. Μου ζητάτε το λόγο, βλέπω, ο Ζαν Πολ. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση μόνο, κύριε Σιγητά, για, το... για την τροπολογία 36 του κυρίου Σμιτ. Λέμε στα γαλλικά, στα γαλλικά υπάρχει ανακολουθία ανάμεσα σε αυτά που... 36, 36. Έτσι, ε, αυτή που αναφέρατε τώρα. Ανακολουθία ανάμεσα στο αν χρειάζεται, αν συντρέχει ανάγκη, αλλά και την αιτιολόγηση όπου λέει ότι για να λειτουργήσει αριθματοσύστημα, το σύστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει οπωσδήποτε να προσφέρει την υποστηρίξη και την τεχνογνωσία τη. Δεν ξέρω στι υπόλοιπε γλωσσικέ εκδοχέ ε, πώ ε, είναι το κείμενο, αλλά στα γαλλικά σαφώ δεν ταιριάζει η τροπολογία με την αιτιολόγηση τη ε, τροπολογία. Γιατί εγώ θεωρώ και μπορεί να μας το επεξηγήσει ο κύριος Σμιτ ότι υπάρχει πράγματι μία ανακολουθία, γιατί αν υπάρχει μία εύλογη συνεργασία, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η Κομισιόν θεωρεί αναγκαίο να παρέμβει. Η τροπολογία λέει ότι αν συντρέξει λόγος θα παρέμβει η Επιτροπή και θα διαθέσει τα κράτη-μέλη κλπ. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που ερμηνεύει. Ποιος είναι ο υποκείμενος ε, ερμηνείας. Βεβαίως ίσως ο κύριος Σμιτ μπορεί να μας την ε, επεξηγήσει και μπορεί να μας πει μέσα στη, στα πλαίσια της οξυδέρκειας που τον διακρίνει περί τι ακριβώς περί πρόκειται. Όλα. Ο κύριος Μαγκάλο βρήκε σωστή ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα στοιχεία που πρέπει να καλύπτει η έκθεση. Δεν νομίζω να διαφωνούμε σε τέτοιο βαθμό. Και συμφωνώ με την τροπολογία 28 με την αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την πελώρια πάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Τώρα για τις υπόλοιπες τροπολογίες είμαι φιλελεύθερος, έτσι. Λέτε εσείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί, καν. Εγώ λέω shall ή should, θα ή θα έπρεπε. Καταλαβαίνετε, εγώ ακολουθώ τη μέση εδώ. Και προσθέτω, if necessary, αν συντρέχει ανάγκη. Αν μπορείτε να δεχτείτε shall, αυτή τη διατύπωση, θα συμφωνήσω μαζί σας. Έτσι θα ευθυγραμμιστούν περισσότερο οι θέσεις μας. Είχα μπερδευτεί, ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, λέει ο κύριος Μαργκάγιο, για τη συνεργασία τους και ε, εάν ε, εκείνοι που έχουν ε, προβάλλει τροπολογίες θέλουν να μιλήσουν μαζί μου, είμαι στη διάθεσή τους, όποτε το θελήσουν. Και άλλοι θέλουν το λόγο. Ούντο, πρέπει να μιλήσεις, ντε και καλά, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εξ ονόματο τη Κάθριν Στήλερ, η οποία είναι σκιώδη, θα ήθελα να σας πω ότι υποστηρίζει το πνεύμα της έκθεσης και τι τροπολογίε ε, που υποβάλαμε δεν θέλανε να αναιρέσουν την έκθεση, να την ενισχύσουν ήθελα. Γι' αυτό ελπίζουμε να υποστηρίζετε εσείς εισηγητά της. Ε, Τροπολογίε μα Ολοκλήρωσα λοιπόν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου δώσατε. Μάλιστα, έχουμε καθυστερήσει 12 λεπτά γιατί ξεκινήσαμε στις 3 και 12 λέει ο πρόεδρο. Όχι επειδή έλειπα εγώ, επειδή λείπατε εσείς βασικά. Να περάσουμε στο 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 σε όλο το πακέτο για την δέσμη χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Να προτείνω να κάνουμε το εξής. Να ακούσουμε από κάθε έναν από τους εισηγητές 7 το αριθμό τι έχουν να μας πούν και μετά οι σκιώδεις και οι υπόλοιποι να μου ζητήσουν το λόγο και θα τους τον δώσω μετά. Ωραία λοιπόν και πάλι να ακούσουμε για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών τον κύριο Μαργαϊό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα από τα πιο βασικά θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν σε αυτή τη θητεία θητεία νομοθέτησης και είναι και μία από τις μεγάλες προκλήσεις της Ισπανικής Προεδρίας. Θα μιλήσουμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το, τους συστημικούς κινδύνους και να μπορούμε να ελέγξουμε και το, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τη, τους τραπεζικούς φορείς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Διότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη σύμπνοια. Τώρα, για να δούμε πώς ορίζεται αυτό το σύστημα, θεωρώ ότι όλες αυτές οι αρχές θα πρέπει να έχουν μία ενιαία έδρα, τουλάχιστον όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία και τα τραπεζικά ιδρύματα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τους συστημικούς κινδύνους. Δηλαδή να υπάρχει ένας εποπτικός έλεγχος, ιδιαίτερα για καταστάσεις επίγουσας ανάγκης. Εδώ η Επιτροπή θέλει απόλυτο έλεγχο αλλά και το Συμβούλιο ως προς την αντιμετώπιση συστημικού κινδύνου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατεπίγουσα κατάσταση. Ιστορικά, το Κοινοβούλιο ε, δεν λαμβάνει το λόγο επί του θέματος για πρώτη φορά. Θα ήθελα λοιπόν, πριν τροποποιήσουμε αυτές τις εκθέσεις, θα πρέπει να λάβουμε την προγενέστερη έκθεσή μου του 2000 σε σχέση με την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διότι αυτό που έχει σημασία είναι μια στοχοθέτηση, η απελευθέρωση των αγορών, η εποπτεία και ο έλεγχος και η εναρμόνιση του φορολογικού συστήματος. Και πιστεύω ότι όλα αυτά έπρεπε να τα δούμε, θα έπρεπε να τα δούμε με κάποια σπούδη, έτσι ώστε να υπάρξει ένας συγχρονισμός για να μην ανακύψει συστημικός κίνδυνος. Αυτό το έλεγα στην έκθεσή μου του 2000 διότι μιλάμε για ενοποίηση, παγιοποίηση από τη μία πλευρά και εποπτεία από την άλλη. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι η χωροταξική κατανομή των διάφορων χρηματοπιστωτικών. Και βεβαίως το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη συνεργασία. Έχει λοιπόν σημασία, έχουν σημασία η ΙΕΡΑ οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, κρίση η οποία μας απασχολεί ιδιαίτερα τώρα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς που θα πρέπει να την χάνουν ευρωπαϊκής εποπτείας. Τέλος λοιπόν, η δική μου έκθεση προτείνει περισσότερη εποπτεία και περισσότερη Ευρώπη. Αυτή είναι, αυτός είναι ο πυρήνας που διέπει την έκθεσή μου. Η κρίση κατέδειξε ότι χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Αυτό τόνισε και ο νέος επίτροπος και ο προγενέστερος διότι η Επιτροπή ε, ζήτησε τη σύσταση μιας Επιτροπής Σοφών. Και η Επιτροπή αυτή συνέταξε μία έκθεση ελάχιστων προδιαγραφών, όπως την ορίσαμε. Από εκεί ανέκυψε και η έκθεση Λαροζιέρ. Και η έκθεση του Συμβουλίου του 2009 έβαλε ακόμα περισσότερο νερό στο κρασί της αρχικής έκθεσης. Και ο κύριος Γκοζές το προανέφερε αυτό, λέγοντας ότι αυτό το κοινοβούλιο δεν μπορεί να δεχτεί την ενιολογική βάση του Συμβουλίου. Η ειρήνη είναι πάντα δυνατή, όπως έλεγε ένας στρατηγός, αρκεί να υποκύψουμε σε αυτή. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Συμβούλιο μιλά τώρα για περισσότερο συντονισμό, περισσότερη Ευρώπη και ούτε καθεξής ε, δυνάμει της τρέχουσας Προεδρίας. Ποια είναι τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν. Θα πρέπει καταρχήν να αντισταθούμε σε αυτό το status quo, γιατί υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις που ανθίστανται. Δεν θέλουν περισσότερες αρμοδιότητες, να εκχωρήσουν περισσότερες αρμοδιότητες. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια ευρωπαϊκή βίβλο, κοινούς κανόνες, για να ερμηνεύουμε την ενιολογική αυτή βάση ενία. Εμείς θα θέλαμε, λοιπόν, να τονίσουμε το ρόλο της εποπτικής αρχής. Θα πρέπει λοιπόν να, υπάρχει, να, υπάρξουν, να υπάρξει η τεχνική διαβάθμιση και μετά η εποπτεία καθεαυτή. Και αν στη συνέχεια η Επιτροπή δεν δεχτεί μια πρόταση της εποπτικής αρχής και η εποπτική αρχή δεν δεχτεί την πρόταση της ε, Κομισιόν, τότε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα επιλύσουν αυτή τη διαφορά μεταξύ Κομισιόν και ενιαίας εποπτικής αρχής, αν ανακύψει αυτό το σενάριο. Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω το ρόλο του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Ντεβίγκο γνωρίζει πολύ καλά το θέμα αυτό που έχει σημασία είναι η δράση κατεξουσιοδότηση. Και ως προς τις συστάσεις, αυτό που έχει σημασία είναι ποιες συστάσεις, σε ποιες συστάσεις θα προβούμε. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για υποχρεωτικό ή δεσμευτικό πλαίσιο. Υπάρχει και αυτό αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πώς ορίζονται και οι αρμοδιότητες του εκτελεστικού σκέλους, της εκτελεστικής αρχής. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα. Ο αρμόδιος πρόεδρος αυτής της εποπτικής αρχής θα πρέπει να έρθει ενώπιον μας για να δούμε ποια ε, εποπτικά πλαίσια χρειάζονται σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να φτάσουμε σε αίσιο πέρας. Να δούμε δηλαδή τι εκχώρηση κεφαλαίου χρειάζεται από ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα εκεί όπου χρειάζεται. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή μπορεί να ανταποκριθεί στα προαπαιτούμενα που προβάλλει μία έρα, δηλαδή μία εθνική ρυθμιστική αρχή. Ποιε θα είναι δηλαδή οι αρμοδιότητες του Ευρωπαίου επόπτη. Θα πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε εάν υπάρχει το απόλυτο κενό. Ο Γκαρθία Ορτέγκο ε, λέει ότι οι επίπονες προσπάθειες ε, πολλές φορές δεν αποδίδουν. Θα πρέπει να πούμε δηλαδή τι θα γίνει σε περίπτωση παράβασης ή παράληψης δυνάμει της συνθήκης. Επίσης, τι θα γίνει σε, σε περίπτωση κατεπίγουσας ανάγκης με βάση συστημικό κίνδυνο και τι θα γίνει αν υπάρχει ανακολουθία μεταξύ ΕΡΑ, δηλαδή Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών και Ευρωπαίου Επόπτη. Εμείς εδώ βάζουμε προθεσμίες ενισχύουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου, το δημοκρατικό έλεγχο για να αντιμετωπίσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα και να δώσουμε, να προσδώσουμε μεγαλύτερες αρμοδιότητες στην εποπτική αρχή. Σε αντίθεση με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειαζόμαστε μια πιο ε, δυναμική και ευρωπαϊκή εποπτική αρχή. Εδώ υπάρχει το κεντρικό μας θέμα, το θέμα της εποπτείας. Θα ήθελα να διαβάσετε το Turner Review που σχετίζεται και με την έκθεση Rosière άμεσα. Το Turner Review αναφέρει ότι η κρίση κατέδειξε ότι οι μηχανισμοί που είχαμε θέσει σε εφαρμογή για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν οδήγησε στην αποφυγή της ρήξη του συστήματος. Και λέει ότι υπάρχει ε, το θέμα της Ισλανδίας το οποίο είχε επιπτώσεις και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε μία μητρική επιχείρηση την έδρα δηλαδή, σε σχέση με τις θηγατρικές. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να εποπτεύσουμε το καθεστώς φερεγγιότητας στις ε, θηγατρικές. Γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μία ε, προστατευτική πλαισίωση, κάτι το οποίο δεν θα ήταν σωστό. Αυτό λέει το Turner Review, η επιθεώρηση αυτή. Θα πρέπει να βασιστούμε λοιπόν στο εξής οι εθνικές ε, αρχές, μάλλον τα εθνικά ιδρύματα τα οποία ε, δρούν σε εθνικό επίπεδο δεν έχουν ε, επιπτώσεις προς τα έξω. Αυτό που έχει σημασία είναι τι γίνεται σε περίπτωση διασυνοριακής συνεργασίας ή εκεί όπου υπάρχει έδρα και θηγατρικές. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, τι διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει, δεσμευτική διαμεσαλόβηση, όταν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ εποπτικών αρχών και κατά πόσο μπορούμε να έχουμε άμεσες αποφάσεις τη στιγμή που δεν υπάρχει μία προγενέστερη πλαισίωση. Τρίτον, θεωρώ ότι οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι δεν θέτουν πολλά προαπαιτούμενα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ευρωπαϊκή εποπτεία προς όλα αυτά τα ιδρύματα διαμέσω των ΕΡΑ, των Εθνικών Εποπτικών Αρχών, των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών και των ε, Εθνικών Εποπτικών Αρχών. Γιατί εάν είχε προϋπάρξει κάτι τέτοιο, τότε θα είχε θα, είχαν αντιμετωπιστεί, θα είχε αντιμετωπιστεί πληθώρα κρίσεων. Γιατί έτσι ξέρουμε ποια είναι τα προαπαιτούμενα και πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτό το ε, οικοδόμημα των ε, εποπτικών αρχών, της Ευρωπαϊκής ε, Εποπτικής Αρχής. Εάν λοιπόν η αρχή είναι ευρωπαϊκή, πού είναι, σε ποιον είναι οι υπόλογη αν υπάρξει θεσμική καταβαράθρωση. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να συρρυκνώσουμε τους κινδύνους. Δηλαδή, θα πρέπει. Θα πρέπει να έχουμε ένα ταμείο το οποίο προχρηματοδοτείται από τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές έτσι ώστε να μην υπάρχει διπλή φορολόγηση και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε εγγύηση καταθέσεων και διάσωση καταθέσεων και κατά δεύτερον το Ταμείο όταν δεν έχει αρκετούς πόρους μπορεί να προβάλλει ένα καθεστώς έκδοσης ομολογιών έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Και εάν τα κράτη πρέπει να παρέμβουν, θα ήταν καλύτερα να δράσουν με βάση ένα Memorandum of Understanding παρά να φτάσουμε σε μία κρίση. Εδώ σκέφτομαι τη, Force, τη και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έτσι ώστε να αποτελέσει αυτή η αρχή ένα ανάχωμα και να έχουμε σωστή ρευστότητα στις αγορές και να φυσικά να εγγυηθούμε και τις καταθέσεις. Να υπάρχει μια εγγυοδοσία των καταθέσεων. Αυτή είναι η ενιολογική ε, βάση της έκθεσης. Και τώρα αρχίζει η πραγματική εργασία. Χρειάζεται μεγαλύτερη εποπτεία, περισσότερη Ευρώπη και λιγότερος κίνδυνος για τους φορολογούμενους. Αυτές είναι οι τρεις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν αυτή την έκθεση και πιστεύω ότι αυτή θα είναι η πραγματική συνεισφορά μας, όπως όρισε και η Ελίζα Φερέιρα. Γιατί πιστεύω ότι με βάση αυτή την ιβυρική συνεργασία θα φτάσουμε να αγγίξουμε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Um, uh, Ευχαριστώ. Ο Σβέν Γκίγκολντ ε, τώρα, εισηγητής ε, για τις ε, αρχές, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι πέρα από την Ισπανοπορτογαλική φιλία ελπίζω και στο θέμα αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο να δημιουργήσουμε μια φιλία, αν θέλετε, μεταξύ Βορρά, Νότου, Ανατολής και Δύσης της Ευρώπης. Γιατί δεν επικρατεί πάντα ομοφωνία σήμερα μεταξύ του τι γίνεται στην κεντρική βόρεια-νότια ε, Ευρώπη. Και εδώ, στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να δώσουμε την απάντηση αυτή στην κρίση, όπως είπε ο συνάδελφος Μαγκάγιο. Να πούμε δηλαδή ότι η απάντηση στις προφανείς ελλείψεις ε, κοινών κανόνων και κοινή δράσης να αντιμετωπιστούν σε πλαίσιο α, νομισματικής πολιτικής αλλά και οικονομικής πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την επέκταση, τη διεύρυνση τη συνεργασία, όχι με τον περιορισμό τη συνεργασία μα, γιατί αυτό θα αποτελούσε ασφαλμένη απάντηση στην κρίση. Και γι' αυτό χαιρόμαστε που ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι ε, δομέ εποπτεία, όχι μόνο των τριών ε, εμ, ε, ιδρυμάτων αυτών, αλλά και σε γενικότερο επίπεδο να δοθεί μια τριθωτική απάντηση σε ό,τι αφορά την χρηματοοικονομική εποπτεία και την αντιμετώπιση της ε, κρίσης στον τομέα της, ε, του συστημικού κινδύνου. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω όσα ήδη έχουμε ακούσει απλά και μόνο επειδή αναφέρονται στην έκθεσή μας. Μόνο ορισμένα σημεία θα ήθελα να θίξω. που ίσως να υπάρχει μια λεπτή διάκριση μεταξύ των ε, εκθέσεών μας. Γιατί οι δύο εκθέσεις ε, είναι πολύ παρόμοιες. Είμαστε επιπισμένοι ότι τα μεγάλα διασυνοριακά ιδρύματα θα πρέπει να υπόκεινται σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και φυσικά λογικό στην επακόλουθο είναι ότι θα πρέπει να δοθεί και μία απάντηση για το ποιος πρέπει να πληρώσει όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Δεν είναι δυνατόν να είναι τα κράτη-μέλη αυτά, τα οποία θα πληρώσουν αν δεν ήταν τα υπεύθυνα εποπτείας. Κάτι άλλο. Για το ποιος πληρώνει και πάλι και ποιος πλήττεται από τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπο, όπου το ίδιο πνεύμα διέπει και τις τρεις εκθέσεις. Είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν μπορεί να επιτρέπεται στο άρθρο 23 να αναφέρεται απλά ότι ναι, αν υπάρχει αντίκτυπος, οποιοδήποτε αντίκτυπος στα δημοσιονομικά των κρατών μελών υπάρχει δικαίωμα βέτο, άρνηση κυρίας, αυτό θα οδηγούσε σε έναν παραλογισμό την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή επειδή πρέπει να μετακινηθούν κάποιοι υπάλληλοι, αυτό έχει αντικτύπω στα δημοσιονομικά των κρατών μελών. Δεν μπορεί να είναι αυτό ο στόχο μα και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα παράλογο. Είναι πραγματικά πολιτική κομμωδία να αποστέλνουμε επιστολή στο Συμβούλιο και να ρωτάμε αναφορικά με την πρωτοβουλία του Πίτερ Σκίνερ και να ρωτάμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη και να λαμβάνουμε ως απάντηση ότι «Α, ξέρουμε ότι είναι δύσκολος όρος αυτός, ευχαρίστως να το συζητήσουμε μαζί σας». Δεν γίνεται έτσι η νομοθεσία, λυπάμαι. Είναι κομμωδία αυτό. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε στο σημείο αυτό να αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αποδείξουν ότι μια ευρωπαϊκή απόφαση επηρεάζει όντω τον, τον προπολογισμό τους, ιδάλλως δεν υπάρχει λόγος να τίθενται ευρωπαϊκοί κανόνες. Ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρώ είναι σημαντικό για τον τομέα τον οποίο χρειάστηκε να εξετάσω εγώ για τη νέα Ευρωπαϊκή Αρχή που θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αναφορικά με συγκεκριμένα προϊόντα να τα αποκλείει από την αγορά. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου για παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι απαγορεύονται η κερδοσκοπία με, ε, με τα κρατικά ομόλογα της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να έχουν οι ευρωπαϊκές αρχές, γιατί πλέον έχουμε μάθει ότι υπάρχουν εν μέρη δραστηριότητες στην αγορά που θα πρέπει που δεν σχετίζονται απαραίτητα με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και αυτό προβλέπεται στην έκθεσή μου. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα επίσης να συζητήσω περαιτέρω μαζί σας είναι το θέμα του Board of Appeal. θεωρούμε ότι αυτή η κοινή επιτροπή θα πρέπει να ενισχυθεί και δεν είναι μυστικό. Και ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι με παρόμοια άποψη εδώ ότι δεν είναι πολύ λογικό αυτό. Δεν είναι λογικό να υπάρχουν τρεις διαφορετικές αρχές οι οποίες να πραγματεύονται ουσιαστικά παρόμοια, παρόμοιες αγορές. Ούτε να έχουν έδρα σε τρεις διαφορετικές πόλεις. Είναι λογικό. Αυτό σημαίνει ότι σε περιπτώσεις ε, κρίσης δεν υπάρχει ουσιαστικά τόσο πολύ ανεπίσημη επικοινωνία. Επικρατούν τρεις διαφορετικές κουλτούρες και το καθεξής. Η ενίσχυση της κοινή επιτροπής αποτελεί έναν τρόπο για να κινηθούμε προς την κατεύθυνση τουλάχιστον μιας κοινή υποπτικής αρχής και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε στην Επιτροπή μας το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το κοινό με ακριβώς, προκειμένου τελικά να καταλήξουμε σε μια ενοποιημένη Ευρωπαϊκή Υποπτική Αρχή. Οι εκθέσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Και από ό,τι μας έχει διδάξει και η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι οι στόχοι που διατυπώνουμε δεν θα πρέπει να είναι θεωρητικοί, θα πρέπει να έχουν ε, ως ε, στόχο την επίλυση των προβλημάτων. Αν παραμείνουμε σε αυτό το θεωρητικό επίπεδο, δεν θα πετύχουμε τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά φυσικά, να μην ξεχάσουμε και τις βασικούς κανόνες που αναφέρονται για παράδειγμα στο Ντελόρ. Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα και από κοινού να προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού να πραγματοποιήσουμε το βήμα αυτό. Ε, ε, Σας ευχαριστώ και τώρα να περάσουμε στην έκθεση του Πίτερ Σκίνερ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Ο Πίτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ενδιαφέρουσες. Ε, συζητάμε αυτά τα θέματα και σίγουρα όλοι θέλουν να εξασφαλίσουν το αποτέλεσμα θα είναι χρήσιμο ε, για τις συζητήσεις μας με το Συμβούλιο, αλλά να έχει και κάποιο όραμα. Δηλαδή να έχουμε επίγνωση όχι μόνο το τι χρειάζεται για τις επιχειρήσεις, αλλά να ικανοποιήσουμε τους κατάλλοντες και τους πολίτες της Ένωσης. γιατί τώρα αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και των ρυθμιστικών αρχών. Γι' αυτό συνέταξα μία έκθεση για την εξυγίανση και την ενσωμάτωση στον κλάδο Δέχομαι το πνεύμα της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όμως πιστεύω ότι χρειάζεται ένα σύστημα ελέγχου ε, που ίσως γνωρίζετε. Ε, κάτι δηλαδή που θα περίμενε κανείς από μια έκθεση του Κοινοβουλίου. Σε τι διαφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δίνει το ρυθμό, όπως είπε ο Χωζε Μανουέλ. Θέλουμε κάτι που να ικανοποιεί το Κοινοβούλιο, όχι αυτό που θέλει να μας σερβίρει το Συμβούλιο. Εμείς θέλουμε να θέσουμε τους όρους ισότιμα με το Συμβούλιο. Έχω έξι βασικά ζητήματα. Σύντομα θα τα διατρέξω για να καταλάβετε το γενικότερο πνεύμα των συζητήσεων που έχουν προηγηθεί. Και εξαλλού θα ήθελα ενδεχομένω να προσθέσω και άλλα σημεία, σημεία που θέλω να συζητήσω με του συναδέλφου μου. Πάντω υπάρχει ευρεία συνένεση. Επιπρόσθετε αρμοδιότητε για το Κοινοβούλιο, για τον έλεγχο, ε, ε, κατάργηση κάποιων αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ευθύνη, στη ρήτρα διαφύληξης, καλύτερη νομοθεσία, όλα αυτά ε, συνιστούν ένα πλαίσιο για την χρηματοπιστωτική εποπτεία και μια μεικτή επιτροπή και ε, επίση ε, βασικό ρόλο κάποιων εξωτερικών παραγόντων. Και δίνω για συγκεκριμένα παραδείγματα, ούτω ώστε ε, να μπορέσω να πάρω την υποστήριξη από του συναδέλφου μου. Επιπρόσθετε αρμοδιότητε για το Κοινοβούλιο. Όλοι συμφωνούν. Θα επιλέγουμε του προέδρου του, από κάποιου τελικού καταλόγου για όλε αυτέ τι αρχέ και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Η επικεφαλή των αρχών θα υποβάλουν τα πρακτικά εκθέσεις ε, στο Κοινοβούλιο και θα μα δίνουν πρόσθετε πληροφορίε όταν εμεί τι χρειαζόμαστε, όχι όταν εκείνοι αποφασίζουν ότι πρέπει να έρθουν σε επαφή με το Κοινοβούλιο και ορισμένε φορέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντάξει το λέω λίγο ομά, ε, θέλει όλο ένα και περισσότερε αρμοδιότητες και θέλει εκείνη να διορίζει όλου του επικεφαλεί των αρχών και τη μορφή των εκθέσεων που μα ε, υποβάλλει. Ε, θα πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε ηγετικό ρόλο. Τώρα, κατάργηση κάποιων αρμοδιοτήτων ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, δηλαδή η ρήτρα Omnibus. Ε, ε, θα συμφωνήσω με τον συνάδελφό μου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να τροποποιεί τα τεχνικά πρότυπα, μόνο να, τις εγκρίνει, να τα εγκρίνει μπορεί εν μέρη ή πλήρωση, να τα καταργεί. Αυτό πρέπει να είναι το πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ESRB τώρα, όπως είπε ο κύριος Μαργές, ε, και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κρούσει τον κόδωνα ε, του κινδύνου ότι είναι πήγουσα η κατάσταση. Δικό τη ρόλο είναι ο Σβέν. Ε, είπε κάτι πολύ εύστοχο. Η επιστολή που στείλαμε και που απερίφθη από το Συμβούλιο χωρί καμία εξέταση, πρέπει να το πούμε, είναι χαρακτηριστική. Υπάρχει αυτή η ρήτρα διαφύλαξη για την δημοσιονομική ευθύνη, fiscal responsibility. Μα τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορεί να το αφήσουμε στα χέρια χέρια ενό δημοσίου υπαλλήλου που τα λέει με ένα δημόσιο υπάλληλο σε μια άλλη χώρα. Δεν είναι αυτό ευθύνη. Πρέπει να έχουμε αξιολόγηση αντικτύπου, να έχουμε περιγραφή μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά όλοι τι αρμοδιότητέ μα και το Συμβούλιο. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που να μα βολεύει και εμά. Καλύτερη νομοθεσία λοιπόν. Τι απαιτείται, Αξιολόγηση αντικτύπου. Ε, αυτά που ζητάμε εμεί είναι να καταλάβουμε καλύτερα το πώ λειτουργούν τα τεχνικά πρώτα και πώ εκδίδονται οι τεχνικέ σε κατευθυντήριε ε, γραμμέ, να μην βασιζόμαστε μόνο στι βέλτιστε πρακτικέ, ε, να βρίσκουμε πιο λογικού τρόπου για να αποφασίζουμε. Τώρα, μεγαλύτερη ενσωμάτωση και καλύτερη εξυγίανση. Το ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας μπορεί να το φροντίσει αυτό και να υπάρχει σαφής ρόλος για την Ευρωπαϊκή Αρχή, την ESRB. Ε, τώρα, ε, ο ρόλος της Μικτής Επιτροπής ε, πρέπει να αποαχθεί ούτως ώστε να αποτελέσει βάση για μια πιο εν, ολοκληρωμένη ένα πιο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό εποπτικό σύστημα. Αυτό χρειαζόμαστε, διότι δεν αρκούν οι αρχές. Ξέρετε όλοι ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ημών και ημών για να ε, δούμε ακριβώς αυτό που ε, κυοφορούμε τώρα σε τι θα οδηγήσει. Αλλά ο Χωζέ Μανουέλος Βεν ε, δεν το έχουν συζητήσει αυτό μαζί μου αλλά δείτε στην έκθεσή μου τις μελλοντικέ προοπτικές όπως τις προδιαγράφω για να μιλήσουμε όλοι με μία φωνή. Έκτον, ε, υψηλότερη εκπροσώπηση από εξωτερικού εμπειρογνώμονε. Υπάρχουν ευέλικτε πρακτικέ, αλλά δεν επαρκούν. Ακαδημαϊκοί θα πρέπει να ε, ε, συμμετέχουν στι ομάδε εμπλεκόμενων φορέων και χρειαζόμαστε και νομικούς για να μην έχουμε μόνο τις νομικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει να διευρυνθεί η σύνθεσή του και να μεριμνήσουμε ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να κάνουν αυτό που πρέπει για μας του πολίτε, όχι μόνο για τα όργανα για τα οποία εργάζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πίτερ ε, για το Συμβούλιο Εποπτείας η Σιλβή. Όπως ξέρετε συνεργαστήκαμε όλοι οι προηγούμενοι εισηγητές και οι επόμενοι σε σχέση με τον Γενικό Νόμο Omnibus, την Οδηγία Omnibus. Τρεις κατευθυντήριες γραμμές επελέγησαν για το μακροοικονομικό επίπεδο. Η πρώτη προελέχθη, δηλαδή να προσεγγίσουμε το μάκρο και μικροοικονομικό ε, επίπεδο καθώς και τις μάκρο και μικροοικονομικές αναλύσεις διότι οι κυβερνήσεις που θέλουν ξεχωριστές οντότητες δεν μας δώσαν πιστικά στοιχεία. Δηλαδή διανύζουμε ένα σχήμα. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να περάσουμε, να κάνουμε ένα ουσιώδες βήμα, όπως είπε και ένας προλαλή σας. Θα πρέπει να έχουμε μία κοινή εποπτεία, κοινή εποπτική βάση. Αυτό ελέγχθηκε στις ε, ακροάσεις και, στην, και από την έκθεση Λαροζιέρ, τονίστηκε. Θέλουμε ένα μακρόπνο σχέδιο έτσι ώστε να έχουμε κάθε ευκαιρία. Εκεί όπου δεν υπάρχει εμπιστοσύνη να υπάρξει λίγη περισσότερη και να έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Θα θέλαμε το μέλλον να παραμείνει ανοιχτό προς ε, μια πορεία ολοκλήρωσης εάν το κρίνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μετά από ορισμένα χρόνια. Η δεύτερη ανησυχία έγκυται στο εξή. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τα κατάλληλα μέσα και όργανα που χρειαζόμαστε. Συνολικά. Επιμένω σε αυτό. Γιατί αν δούμε τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο, στη ΣΥΠΑ δηλαδή, βλέπουμε ότι κανείς δεν έχει την ε, ιδεατή λύση υπάρχει ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός έτσι ώστε να ορίσουμε νέους κανόνες. Και αν δεν είμαστε παρόντες ως Ευρώπη, οι αποφάσεις θα ληφθούν αλλού. Άρα στην έκθεση αυτή θέλω να διασαφηνίσω ένα σημείο. Η Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου βρίσκεται υπό την ΕΤΕ και η έκθεση Λαροζιέρ ορίζει ότι ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας θα είναι ο πρόεδρος. Θα πρέπει λοιπόν να, υπάρχει, να έχουμε να κάνουμε με μια δυνατή και δυναμική αρχή έτσι ώστε να μην χρυσώσουμε το χάπι. Ο πρόεδρος αυτής της Ευρωπαϊκής Αρχής θα είναι υπεύθυνο ε, για την Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο και θα πρέπει να το διασφαλίσουμε ενώπιον των Ευρωπαίων, να μην κρυβόμαστε γιατί αν γίνει ε, μία εκλογή σε επίπεδο κεντρικής τράπεζας, ίσως χάσει την εκλογή αυτή ο πρόεδρος, ο διοικητής. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τις ε, αρμοδιότητες, δηλαδή την λογοδοσία αυτού του οργάνου ενώπιον Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπως είπε και ο Πίτερ Σκίνερ θα υπάρχει αυξανόμενος έλεγχος στις μικροοικονομικές αρχές. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα έρχεται ενώπιόν μας για την αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου. Θα υπάρξει μια διαδικασία πρόληψης και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει λογοδοσία και δικαιοδοσία. Άρα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα βρίσκεται υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα πρέπει η υπεύθυνη της εποπτείας, είτε πρόκειται για διοικητές κεντρικών τραπεζών ή υπουργών οικονομικών ή αν έχουμε μία πρόσμιξη των δύο, θα πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μία κρίση. Έτσι ώστε και αν ανακύψει κρίση να μπορέσουμε να ε, λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα σε επίπεδο Συμβουλίου Συστημικού Κινδύου. Κινδύνου. Να μην έχουμε εκπροσώπους λόμπι ή συγκεκριμένων αρχών, αλλά αυτόνομες προσωπικότητες που να μπορούν να εισαγάγουν ε, στοιχεία, λυσιτελή στοιχεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Επίσης, το προσχέδιο της Επιτροπής προέβλεπε μια τεχνικής ε, υφής επιτροπή ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων. Εγώ τονίζω ότι η Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου μπορεί να λάβει υπόψη και αρμοδιότητες εποπτικής αρχής ή των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Θα πρέπει όμως να έχουμε ακαδημαϊκούς ε, του υψηλότερου δυνατού επίπεδου από παντού ε, ανά τον κόσμο. Δεν δίνουμε απάντηση σε όλα τα στοιχεία. Θελήσαμε όμως να ανοίξουμε μια συζήτηση έτσι ώστε ορισμένα λόμπι οι κυβερνήσεις να μην γυρίσουν στην αρχή του business as usual. Πρόκειται για ένα συλλογικό εγχείρημα. Ίσως υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε τις γενικές αρχές και πιστεύω ότι σε αυτούς τους γενικούς ενιαίους κανόνες να είμαστε πιο δυνατοί ενώπιον του Συμβουλίου. Γιατί έχουμε εκλογικές περιφέρειες όπου βλέπουμε τους συμπολίτε μας να αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας, να έχουμε Ε που αντιμετωπίζουν μια μεγάλη κρίση και και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν άλλαξε τίποτα. Ευχαριστούμε. Τώρα θα ασχοληθούμε με τα ειδικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ο Ραμόν έχει το λόγο. Η έκθεση μου είναι πολύ σύντομη συνέγραψα αυτή τη μικρή έκθεση όπου προβλέπω ε, μια αιτιώδη συνάφεια, έναν ειδικό δεσμό δηλαδή μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να είναι και πρόεδρος του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, έχει ολοένα και μεγαλύτερη αξιοπιστία τη τελευταία δεκαετία και θεωρώ ότι πρόκειται για ένα όργανο το οποίο έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο και πολλοί Αγγλοσάξονες το, αντίπισαν, το, ανέφεραν αυτό όπως ο David March ο οποίος είναι επικριτικός αλλά θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κέρδισε μεγάλη αξιοπιστία τα τελευταία δέκα χρόνια. Θα ήθελα να το συζητήσω με τους Αγγλοσάξονες εάν πιστεύουν ότι υπάρχει αυτός ο ειδικό δεσμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο μόνος ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας ή όργανο που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή, επί της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής που χρειαζόμαστε. Άρα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να παρουσιάζει στο Συμβούλιο του Συστημικούς Κινδύνους και θα ήθελα να υποβάλω μια τροπολογία στο κείμενο έτσι ώστε ο πρόεδρος, που τώρα είναι ο κύριος Τρίσε, να εμφανίζεται ενώπιον του Κοινοβουλίου σε τακτά ε, χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ενώπιον των πολιτών για να ξέρουμε πώς ε, διαχειριζόμαστε την κρίση. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει στη Γενική Γραμματεία να δίνει όλα τα στοιχεία και την ε, διοικητική και επιμελητιακή στήριξη. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να χρηματοδοτεί η ίδια το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Τέλος, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συστημικού Κίνδυνου θα είναι ο οργανισμός που θα διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών σε μικρο και μακροοικονομικό επίπεδο και αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, γι' αυτό θα πρέπει να ισχύει η ρήτρα απορρίτου ή εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ πολύ, με χαρά θα δεχτώ τα σχόλιά σας και τις υποδείξεις σας. Um, Τώρα προχωρούμε στο Omnibus 1. δηλαδή οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Ο Αντολίν Σάντσες Πρεζέδο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω μόνο στα πλαίσια του Omnibus 1. Η οδηγία Omnibus 1, η γενική οδηγία Omnibus 1, θέλει να ανασκευάσει τις 11 τομεακές οδηγίες που διέπουν τον τραπεζικό τομέα και τις κινητές αξίες έτσι ώστε να επαχθούν στο νέο ευρωπαϊκό εποπτικό σύστημα. Αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας αφορά τρεις αρχές σε επίπεδο μικροεποπτείας. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κατακαιρματισμένο σύστημα όπου συνεργάζονταν οι εθνικές εποπτικές αρχές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση. Στόχος είναι να ενταχθούν αυτές οι αρχές στο σύνολο των οδογιών να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ παλών και νέων αρχών, να οριστούν διαδικασίες έτσι ώστε να ρέουν οι πληροφορίες μεταξύ αυτών των αρχών και επίσης η διασφάλιση οδηγιών ή κατεξουσιοδότηση πράξεων. Επίσης, εποπτικές πράξεις και μια γενικότερη, ένας γενικότερος συντονισμός μέσα από διευθυντικά όργανα. Πρόκειται για έναν συντονισμό που είναι καθαρά τομεακός και θα πρέπει να είναι και δύο συνοριακός όπως θα ορίζει η Joint Committee. Τα ζητήματα αυτά δεν αφορούν επικαιροποίηση των οδηγιών που προϋπάρχουν, αλλά αναθεώρηση των οδηγιών, έτσι ώστε να ενσωματώσουμε τις τροποποιήσεις εποπτικής ε, υφής για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και υπάρχουν δύο σημαντικές ε, πτυχές εδώ. Καταρχήν, η αλλαγή πλαισίωσης πορίζει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Στο άρθρο 260 μιλάμε ε, για κατεξουσιοδότηση πράξης και στο άρθρο 291 η συνθήκη αναφέρει τις εκτελεστικές πράξεις. Υπάρχει και διαδικασία Λαμφαλούζη όπου ορίζει ε, μία νομοθετική αρχή σε πρωτογενές επίπεδο. Τώρα όμως διευρύνουμε το πλαίσιο με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 290. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι αυτές και ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που εντάσσονται είτε στις ε, εκτελεστικές πράξεις είτε στις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ενσωματωθούν στις ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση. Οι άλλες ε, διατάξεις θα πρέπει να αξιολογηθούν διότι δεν πρόκειται για την αρχιτεκτονική λαμφαλούση, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή βάση εποπτείας. Και αυτό σημαίνει εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα δεν εφαρμόζουμε απλώς, αλλά λέμε μέχρι που εναρμονίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό θα αφορά τις πράξεις εξουσιοδότηση κατά προτεραιότητα, έτσι ώστε να βρεθούν και οι εκτελεστικές πράξεις κατά συνέπεια. Το Single Rule Book αφορά μία ενιαία βίβλο. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο, διότι η Κομισιόν δεν ταξινόμησε ούτε όρισε τις αναπτυξιακές δράσεις νομοθετικού περιεχομένου. Θα πρέπει λοιπόν να διακρίνουμε τρεις πτυχές στα πλαίσια του Single Rule Book όταν πρόκειται για ορισμούς θα πρέπει να έχουμε κοινού ορισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι εθνικές οντότητες να έχουν κοινού κανόνες ε, ε, παιχνιδιού. Επίσης, οι τεχνικές reporting και αποκαλύψεων, disclosure, αφορούν οικονομικούς φορείς αλλά και το κοινό, το οποίο θα πρέπει να ξέρει περί τίνος πρόκειται δηλαδή να έχουμε μία ανοιχτή αγορά. Επίσης, μιλάμε για τις διατάξεις που θα διασφαλίσουν τον συντονισμό ε, όλων των οντοτήτων του συστήματος, δηλαδή την υποστηρικτική αρχή μεταξύ εθνικών αρχών. Μιλάμε λοιπόν για ορισμούς reporting και αποκαλύψεις, reporting and disclosure και θεωρώ ότι όλα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει έλεγχος του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπάρχουν 369 τροπολογίες με βάση αυτά τα κριτήρια. Επίσης υπάρχουν τεχνικά standards που δεν αφορούν ε, το MIFID, τη διαφάνεια και ούτω καθεξής. Πρόκειται για πράξεις καθαρά εκτελιστικές, οι οποίες διέπονται από μια συγκεκριμένη πλαισίωση. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι η διαδικασία της επιτροπολογίας δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Άρα εισαγάγουμε τις νέες οντότητες αυτές τις οδηγίες με βάση τα κριτήρια τα οποία σας προανέφερα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπάλτς. Σάντσες, δεν έχει σβήσει το μικρόφωνο σου. Ο κύριος ε, Μπάλτσε δεν θέλει να γίνει άλλη ανταλλαγή απόψεων για το Omnibus 2. Σωστά. Θέλετε να πείτε παρόλα αυτά κάποια πράγματα. Πορά μπορώ να πω, αλλά δεν μπορώ να τοποθετηθώ φυσικά σε ένα, για ένα τέτοιο ανεπίσημο έγγραφο, το οποίο δεν έχω δει ακόμα σήμερα. Η Κομισιόν μίλησε ε, και έθεσε στόχο του τον Απρίλιο, άρα νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε σε κάποια μετέπειτα χρονική στιγμή. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και τώρα να περάσουμε στους κοιόδης εισηγητές και στους υπόλοιπου ομιλητέ. να α, δώσω την το λόγο στους σκιώδες με σειρά που το ζήτησαν. Καταρχάς η Βίκη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους εισηγητές για τις σημαντικές ε, δουλειές που κάναν. Τη σημαντική δουλειά που έκαναν. Η βασική αρχή εδώ είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος στο χρηματοοικονομικό κλάδο σε όλη την Ευρώπη. Και χρειάζονται τρία πράγματα. Σαφήνεια στην εποπτεία της νομοθεσίας, συνοχή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και αντιμετώπιση των κρίσεων, προκειμένου να υπάρχει μια εφικτή διαδικασία που δεν θα ε, επιτείνει, αν θέλετε, τη συγγύηση σε μια κρίση όπως την προηγούμενη. Συμφωνώ με, την, με τον εισηγητή για, ε, το EBA ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα, ίσως το πιο σημαντικό. Το θέμα είναι να ε, υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με διαφανή και συνεκτικό τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Πρώτο περάσω στα θετικά και τα αρνητικά. Θεωρώ ότι είναι κρίμα που δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με τον τρόπο που θα έπρεπε εκτός της ομάδας του εισηγητή. Και ως κοιόδης πρέπει να πω ότι είναι κρίμα που δεν έγιναν συναντήσεις όπως έχουν γίνει για άλλα έγγραφα Επίσης, ε, ο εισηγητής ε, είχε τέσσερις εβδομάδες να υποβάλει τροπολογίες. Εμείς είχαμε μόνο δύο εβδομάδες και ίσως καλό θα ήταν να είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο. Λίγες μέρες παραπάνω ζητώ. Επίσης, στην επιστολή που οι τρεις εισηγητές απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλό θα ήταν να τη δούμε. Όπως και καλό θα ήταν να δούμε και τις απαντήσεις της Επιτροπής. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη να υπάρχει ενιαίος κώδικας και με την ανάγκη να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και καλωσορίζω κάποιες από τις τροπολογίες που υπευλήθησαν. Οι διαβουλεύσεις με την βιομηχανία και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, η διευκρίνηση των, ε, του ρόλου των αρχών σε ό,τι αφορά την εποπτεία, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το καθεξής. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα με το σημείο που θίξατε για την ε, ρήτρα διαφύλαξης, οικονομικής, χρηματοοικονομικής διαφύλαξης. Είχα υπόψη μου κάποιες συμβάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να συνάπτονται ε, με ευκολία, αν θέλετε, αλλά αυτή η ρήτρα διαφύλαξη είναι σημαντική. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παίρνουμε ε, ελαφριά. Είναι σημαντική αυτή η ρήτρα η χρηματοοικονομική. Είναι απόλυτα απαραίτητη γιατί αυτή προστατεύει τους φορολογούμενους που καλούμαστε να προστατεύσουμε και τελικά το άτομο που λαμβάνει την απόφαση για οποιαδήποτε κρίση θα πρέπει να είναι αυτός που πληρώνει τελικά τα σπασμένα, το λογαριασμό. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει ελαφριά να τα παίρνουμε όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε σε ό,τι αφορά την συνοριακή εποπτεία ίσως να μας έχουν βάλει λόγια στο στόμα, γιατί εννοείται ότι χρειάζεται καλύτερη διασυνοριακή παρακολούθηση και εποπτεία. Ωστόσο αυτό θα πρέπει να γίνει με μια πολύ σαφή νομική βάση και κάποια από τις, κάποιες από τις διατυπώσεις που εμφανίζονται στο EBA και στην ΕΣΜΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν νομική σύγχυση. Για παράδειγμα, τότε αναφέρουμε ότι οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να είσαι σε θέση να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες της εταιρεία. Οι οδηγίες, από ό,τι ξέρω, δεν είναι ανομικά δεσμευτικέ για τις εταιρείε, μόνο για τα κράτη-μέλη. Αυτή η νομική λοιπόν αβεβαιότητα θα πρέπει να διευκρινιστεί. Επίσης, για τις εποπτικές αρχές, κατά πόσον θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι στην διακριτική της ευχέρεια. Το δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια διακριτική ευχέρεια σε ό,τι αφορά θέματα που άπτονται τη διασυνοριακή ε, νομοθεσία. Οι εταιρείε χρειάζονται μια συνοχή για το ποιο θα είναι ο εποπτικό του ε, αρμόδιο φορέα. Δεν είναι δυνατόν τη μία μέρα να αντιμετωπίζει κανεί έναν εποπτικό φορέα και την άλλη ε, διαφορετικών. Το θέμα επίσης είναι κατά πόσο υπάρχει το προσωπικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρξει τέτοια εποπτεία για τέτοιε περίπλοκες εταιρείε. Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι όπου λειτουργεί σωστά η εποπτεία θα πρέπει να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των εταιριών και των εποπτών και θα πρέπει να υπάρχει και μια σχέση, αν θέλετε, των εποπτών με την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείε θεωρώ ότι το σύστημα των εθνικών ε, εποπτικών αρχών με τις σχετικά με σχετικές επιτροπές είναι ο καλύτερος τρόπος λειτουργίας και πρέπει να υπάρχει μεταξύ να υπάρξει ισορροπία μεταξύ του απόρριτου και της δημοσίευσης συνδεδομένων. Και ε, σημειώνω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, καλείται για τη δημοσιοποίηση πολύ πιο πολύ περισσότερων πληροφοριών. Ωστόσο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, κάποια δεδομένα τα οποία είναι ευαίσθητα. Και όπου οι εταιρείε έχουν ανησυχία για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απόκρυψη στοιχείων και από τη ρυθμιστική αρχή. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό με προβληματίζει. Κάποιες από τις τροπολογίες με προβληματίζουν. Αν δεν υπάρχει στενή σχέση μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και εταιριών, τελικά οι εταιρείε θα μοιράζονται πληροφορίες με κάποιους ρυθμιστές, για παράδειγμα με την εθνική τους αρχή ρύθμισης, αλλά θα υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών σε μικρές χώρες, για παράδειγμα. Θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία. Τέλος. Είμαι πολύ ευγνώμων για το Ταμείο Εξυγίανσης γιατί αναφέροντας τις λέξεις αυτές καταδεικνύεται πόσο περίπλοκο είναι το θέμα αυτό. Συζητούσαμε προηγουμένως ότι αν ακολουθήσουμε το σουηδικό μοντέλο, το ταμείο αυτό θα αναλογεί σε 2,5% του ΑΕΠ. Ο κόσμος λοιπόν θα πρέπει να κατανοήσει πώς λειτουργεί αυτό το ταμείο. Και διαβάζοντας την διατύπωσή σας ανέκυψαν πολλά ερωτηματικά. Είπατε ότι μιλάμε για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία απειλούν την οικονομική σταθερότητα. Ποια είναι αυτά τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πώς τα μετράμε αν είναι μεγάλα ή μικρά. Και ακόμα και αν περιοριστούμε στα μεγάλα ιδρύματα, πώς θα το ορίσουμε αυτό. Αναφέρεται μετά ότι το Ταμείο θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδώσει χρέη. Πώς το κάνει αυτό, είναι δημόσια οντότητα, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να εγγυηθούν και πώς και σε ποιο βαθμό και σε ποιο νόμισμα. Μιλήσατε για την κατανομή των ε, βαρών. Σημαντικό θέμα αυτό, το burden sharing, για τις καταθέσεις. Πώς στις ε, χοντρικές, λιανικές ε, καταθέσεις, για τα ενεργητικά στοιχεία. Πώς επί τρίτων αξιών, επί των ίδιων αξιών ή μήπως βάση εισόδηματο και τι επίπεδο εισοδήματος θα πάρουμε ως βάση για το καθαρό πριν από, την, από τις απώλειες, μετά τις απώλειες. Όλα αυτά είναι ερωτήματα και ίσως να είμαι και λίγο, να υπερβάλλω λίγο θέτοντας τα ερωτήματα αυτά, αλλά είναι δύσκολα ερωτήματα και αφορούν τεράστιο όγκο χρημάτων. Προσωπικά θεωρώ ότι αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα εδώ στο έγγραφο αυτό, ε, κινδυνεύουμε να ετροχιαστεί όλη η συζήτηση για την υποπτική αρχή και να μην καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τα συστήματα αυτά. Θα ήθελα τα θέματα αυτά να αληθούν στη συζήτηση για την εξυγίανση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος Σάντσες. Ζήτησε και πάλι το λόγο. Θέλεις να επανέλθεις για την τραπεζική αρχή, για τις Eh, Το πρώτο που θα ήθελα να κάνω είναι να ευχαριστώ τον κύριο Γκαρθία Μαργκάγιο για την έκθεσή του πρωτίστως, γιατί δεν πρόκειται για ένα μονόλογο που προωθούμε. Η συνομοθέτηση προαπαιτεί ένα διάλογο και νομίζω ότι στο Κοινοβούλιο θα μιλήσουμε με μία σταθερή και στεναρή φωνή. Ο Ομπέρτο έλεγε ότι δεν θα είμαστε ούτε αποκαλυπτικοί ούτε ζηλωτές. Θέλουμε απλώς να είμαστε φιλόδοξοι. Αυτό θέλει να κάνει το Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχει μια διεθνής ε, εποπτεία δηλαδή τα προαπαιτούμενα αυτής. Εμείς θέλουμε να κατέχουμε έναν ηγετικό ρόλο, να βρούμε ένα πιο αξιόπιστο σύστημα ανά τον κόσμο, έτσι ώστε τα χρηματοπιστωτικά να βοηθήσουν μια βιώσιμη μακροχρόνια οικονομία. Μακροχρόνια οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε τέσσερις ε, ε, κατευθύνσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια προληπτική εποπτεία που να ορίζεται από βασικές αρχές, ε, όχι μόνο με βάση τις αρχές της νομιμότητας, αλλά να ακολουθούμε και τις προδιαγραφές της Βασιλείας με βάση την φερεγγιότητα και την ασφάλεια, δηλαδή βασικές αρχές και όχι μόνο νομιμότητα. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στο σύστημα θα πρέπει να εξεύρουμε μία ε, εξισορρόπηση μεταξύ εσωτερικής αγοράς και αρχής επικουρικότητας. Γιατί θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της ε, προληπτικής αποπτίας ενυπάρχει η επικουρικότητα. Και εδώ μιλάω περισσότερο για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Επίσης θα πρέπει να είναι ένα προοδευτικό σύστημα το οποίο να έχει μία δυνατότητα εξελικτικής πορείας. Πρέπει να είναι ένα καθαρά ευρωπαϊκό σύστημα, ένα οριζόντιο σύστημα, το οποίο να άπτεται όλων των χρηματοπιστωτικών αρχών και εποπτικών αρχών. Δεν, πρόκειται για, δεν θα πρόκειται για ένα κλαμπ μεγάλων οντοτήτων. Αυτό θα ήταν ολέθριο σφάλμα. Θα πρέπει να είναι ένα οριζόντιο σύστημα όπου όλες οι αρχές να ενσωματώνονται και να υπάρχει ένας επιμερισμός ευθυνών όπως προαπαιτούν ορισμένες διαδικασίες. Και όπως ισχύει και από τα διευθυντήρια εποπτικών αρχών που προϋπάρχουν στα εθνικά συστήματα. Θα πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, δηλαδή να υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ μάκρο και μικρο εποπτείας, όπως ορίζει η γενική μας αρχιτεκτονική και να υπάρχει ε, μεγαλύτερη ε, ενσωμάτωση όλων των ε, ε, επιχειρησιακών αρχών. Θα πρέπει να υπάρχει προληπτική εποπτεία, δηλαδή τεχνικά πρότυπα, αλλά και νομοθετική πλαισίωση των ε, προαπαιτήσεων εποπτείας. Άρα η όταν, ας πούμε, υπάρχουν, ε, υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση, early warning από τις μακο, μακροεποπτικές αρχές, αυτό θα πρέπει να υπάρχει, ε, αυτό θα πρέπει να έχει και έναν αντίκτυπο σε early tools δηλαδή έγκαιρη εξέβρεση μέσων για την αντιμετώπιση συστημικού κινδύνου. Αυτό αφορά και το ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό μας απασχολούν και οι οντότητες αντιμετώπισης συστημικού κινδύνου. Άρα δεν μιλάμε μόνο για early warnings, για έγκαιρες προειδοποιήσεις, αλλά και για αρχές που θα μπορέσουν να λάβουν μέτρα. Εδώ δεν μιλάω μόνο για τις ε, τραπεζικές αρχές, αλλά και συγκεκριμένες οντότητες που έχουν ε, ειδικέ διαδικασίες reporting και disclosure αποκάλυψης, αποκαλύψεων. Πιστεύω ότι οι αρχές θα πρέπει να είναι πιο αυτόνομες. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε αυτή την αυτονομία και αυτές οι οντότητες θα πρέπει να έχουν έναν ομοιογενή κατάλογο αρμοδιοτήτων, να μην υπάρχει δηλαδή η ετερογένεια που υπάρχει σήμερα και να εστιάζουμε την προσοχή μας σε μια τεχνική εποπτεία και προληπτική εποπτεία. Ως προς αυτά τα κεφάλαια, συμφωνώ με το φιλοσοφικό υπόβαθρο, δεν πρέπει να εξωτερικεύσουμε το κόστος έναντι των φορολογουμένων πρέπει να εσωτερικεύσουμε το κόστος σε πραγματικό χρόνο, γιατί ζούμε μία χρήση μια μια όπου οι χρηματοπιστωτικές αρχές ζητούν βοήθεια. Δεν μπορούμε να τις ε, καταδικάσουμε σε γρήγορο ή αργό θάνατο. Θα πρέπει να κρατήσουμε τους ζωντανούς να κρατήσουμε αυτές τις αρχές ζωντανές και να μην δημιουργήσουμε μεγάλα προβλήματα στην πραγματική οικονομία. Είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δηλαδή, ε, ρήτρα χρηματοπιστωτικής διασφάλισης. Αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει να προβλέψουμε ένα ανοιχτό το σύστημα stakeholders και να μην μιλάμε μόνο για τις μεγάλες οντότητες, αλλά όλες τις οντότητες ανεξαρτήτως μεγέθους και να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός χώρος εποπτείας. Άρα, όχι κατακερματισμένο σύστημα, όχι συγκεντρωτικό, και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι για να ανταποκριθούμε και για να βγούμε από την κρίση η οποία δεν πρέπει να επαναληφθεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Βόρτμαν ευχαριστώ. Η κυρία Βόρτμαν ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα των εισηγητών, την ομάδα των εισηγητών που μας επέβαλε τις προτάσεις αυτές, γιατί φυσικά Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ε, εκθέσεων, αλλά είναι σαφές, ε, σαφές το κόκκινο νήμα, αν θέλετε, που τι συνενώνει. Για την ιστορική αγορά δηλαδή, για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και μετά από την κρίση, πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η ομάδα των εισηγητών ε, εξάγει και τα απαραίτητα συμπεράσματα, γιατί ένα από τα συμπεράσματα είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουμε μαζί, θα πρέπει να να αντιμετωπίσουμε και να απαλλάξουμε τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών από τα εκατομμύρια που έχουν καταβάλει και θα πρέπει να κάνουμε ένα ευρωπαϊκό βήμα. Συμφωνώ με την κυρία Φούρτ. Δεν είναι τόσο απλό να ορίσουμε τέτοια θέματα σε δύο προτάσεις στην νομοθεσία, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να προκαλέσουμε το Συμβούλιο να κάνει το βήμα αυτό και αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και χαίρομαι ότι δεν μιλάμε μόνο για βορρά και νότο, όπως είπε και ο κ. Γκίγο, αλλά μιλάμε και για Ανατολή και Δύση. Όλα αυτά μας δίνουν μια πολύ ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουμε. Ελπίζω λοιπόν να προκαλέσουμε το Συμβούλιο να ξεπεράσει τη σκιά του που φοβάται. Να μπω σε κάποιες λεπτομέρειες τώρα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον συμβιβασμό του Συμβουλίου, γενικότερα το βασικό μου πρόβλημα με το συμβιβασμό αυτού του Συμβουλίου είναι ότι σε διάφορα σημεία στην όλη την πρόταση εισάγονται διαδικασίες ένστασης όπου το κράτος μέλος τελικά, το Συμβούλιο ε, έχουν την τελική λέξη, την τελική, τελευταία κουβέντα. Και η δύναμη ενός επόπτη, ιδιαίτερα σε δύσκολες ε, καταστάσεις, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υποστηρίζω λοιπόν τις προτάσεις των ευρωπαϊκών εισηγητών για την ε, εξουσιοδότηση, την εξουσία, την αρμοδιότητα που θα πρέπει να υπάρχει στις ε, εποπτικές αρχές και σε ό,τι αφορά τα τεχνικά πρότυπα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μέτρα για καταπήγουσες ε, περιπτώσεις. Το άρθρο 10, περιπτώσεις καταπήγουσες ανάγκης. Θεωρώ ότι είναι σωστά όσα ακούσαμε για το συστημικό κίνδυνο και το σχετικό συμβούλιο. Αλλά ανησυχώ κάπως ως και όδηση ότι το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα κυριαρχείται υπερβολικά από τον τραπεζικό τομέα, γιατί υπάρχουν και άλλοι τομείς στον χρηματοοικονομικό κλάδο που θα πρέπει να ακούσει τη φωνή τους. Αυτό λοιπόν το αναφέρω συγκεκριμένα ως πρώτο σημείο. Τρία άλλα σημεία θα ήθελα να αναφέρω για την έκθεση Giggle κυρίως. Ένα σημείο στο οποίο συμφωνώ απόλυτα είναι η ρήτρα χρηματοοικονομικής διαφύλαξης. Έχει διαβρινθεί πάρα πολύ στο συμβιβασμό του Συμβουλίου και λέει η κυρία Φόρτ ότι έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Ε, κυρία Φόρτ, ιδιαίτερα νομίζω ότι ε, θέλουμε να προστατεύσουμε τα κράτη-μέλη και το Ενωμένο Βασίλειο με τη ρήτρα διαφύλαξης αυτή. Και μάλλον αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουν να δεσμευτούν για μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκίγκολκ ότι αυτή η ρήτρα διαφύλαξη θα πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν γίνεται. Να δούμε και η δική μας νομική υπηρεσία τι θα μπορούσε να αποφανθεί για το θέμα αυτό. Δηλαδή τι απαιτείται νομικά βάση της συνθήκης. Ανυπομονώ λοιπόν να ακούσω Ποιε είναι οι ελάχιστε απαιτήσει βάσει τη συνθήκη εφόσον θέλουμε να περιορίσουμε τη διαφύλαξη. Δύο σημεία του συναδέλφου Γκίγκολτ που με προβληματίζουν ωστόσο. Το πρώτο, απαγόρευση συγκεκριμένων προϊόντων. Και τι θέλει ο κύριος Γκίγκολτ να δοθεί στις ΕΖΑ δυνατότητα παρέμβαση στις εθνικές αρχές. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο. Αναρωτιέμαι μήπως αυτό παραπάει ως μέτρο. Το ίδιο ισχύει και για τις διαδικασίες, κοιτώντας και την ε, συνεκτική εφαρμογή του κριτικού δικαίου, θα πρέπει να υπάρχουν και κυρώσεις σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα μέτρα ή συστάσεις των ΕΖΑ. Θα πρέπει να προσφύγουμε στα εθνικά δικαστήρια. Δεν, είναι καλύτερη, δεν υπάρχει κάποια καλύτερη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Και εδώ σημειώνω ερωτηματικό. Δεν είμαι βέβαιη. Τέλος, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να τεθούν επίσης ώρες. Όχι μόνο κατά την κατάρτιση της νομοθεσίας, αλλά και κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας των, των τεχνικών προτύπων. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εξισωθεί με το Συμβούλιο, με τη σημείωση αυτή, επαναλαμβάνω, και με την Επιτροπή, φυσικά και με τη σημείωση ασφαλώς που έκανα στην αρχή ότι θεωρώ ότι στο έγγραφο, στο συμβιβασμό του Συμβουλίου έχουν ε, συμπεριληφθεί πάρα πολλέ διαδικασίε υποβολή ένστατη και εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προ τα πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Και τώρα να περάσω στον κύριο Μέντε Δεβίγκο, ο οποίο είναι εισηγητή τη Επιτροπή ΑΦΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ήταν να εκπονήσει έκθεση για ε, τα τρία σχέδια, μικρο και μακρο- μακροοικονομικά, ε, προβληματίστηκα γιατί είναι βασικό ζήτημα στην οικονομία και ε, πολυσύνθετο. Είδα με ποιο τρόπο, ποια κατεύθυνση μάλλον φαίνεται να ακολουθεί η νομοθεσία. Οι προτάσεις ε, Λαροζιέρη ήταν ελάχιστες, βέβαια ρεαλιστικές και στη συνέχεια έκανε μια αποδυναμωμένη πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ενέκρινε ένα κείμενο που ήταν ακόμη πιο αποδυναμωμένο. Θα συνεχίσουμε κι εμείς ακολουθώντας αυτή τη ρότα. Ετέβη ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας ε, και πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική άγουσα. Έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε, εκπροσωπούμε τους πολίτες ε, και έχουμε ίσες εξουσίες με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, ναι, εκπροσωπεί τα συμφέροντα των κρατών μελών. Αλλά ε, υπάρχει ισοτιμία ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο παρότι εκπροσωπούμε διαφορετικά συμφέροντα. Οφείλουμε να καταλήξουμε σε μία συνένεση με τους εισηγητές και σκιώδες εισηγητές. Είχα αυτές τις ανησυχίες και φαίνεται ότι ε, συμφωνούν και άλλοι συνάδελφοι μαζί μου. Δεν λέει κανείς ε, κάτι διαφορετικό. Χρειαζόμαστε νέο σύστημα, ευρωπαϊκή εποπτεία. Φυσικά μέσα στο πλαίσιο της νέας συνθήκης ε, χρειαζόμαστε ποπτία και για τις αρχές. Ε, θέλουμε να έχουν νόημα και περιεχόμενο οι νέες αρχές ε, που θα συγκροτηθούν. Είναι νομοθέτημα κλειδί και πρέπει να προσέξουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την κατεύθυνση που περιέγραψα. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων δεν ασχοληθήκαμε με τέτοια τα τεχνικά ζητήματα. Έχουμε ένα σχέδιο με συγκεκριμένε τοπολογίε για τι τέσσερι εκθέσει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, διότι σίγουρα τι γνωρίζετε. Κάτι όμως που ήθελα παρόλα αυτά να αναφέρω είναι το εξής. Το πολιτικό μήνυμα από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων προς το Κοινοβούλιο και προς τον έξω κόσμο πρέπει να είναι επικριτικό παρακαλώ όλοι να ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή. Δηλαδή, έχουμε λάβει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θέλουμε να την υπερβούμε. Θέλουμε να είναι σωστή η ρύθμιση που θα γίνει. Ξέρουμε τι προτείνει το Συμβούλιο, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, εμείς τι αισθανόμαστε ότι χρειάζεται στην Ευρώπη, τι χρειάζονται οι πολίτες, τι χρειάζονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τι χρειάζεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Αυτό είναι το καθήκον που πρέπει να φέρουμε σε πέρας για τις ε, μικρο-μακροοικονομικές εκθέσεις. Ε, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Θα σταματήσω εδώ, Πρόεδρε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, αλλά ε, ας ακολουθήσουμε αυτή τη συνένεση που τώρα διαμορφώνεται, γιατί δεν υπάρχει σοβαρή διάσταση απόψεων. Το ζήτημα αυτό είναι βασικό είναι σημαντικό τώρα που αλλάξαμε κατεύθυνση σε σχέση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την κατεύθυνση. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε κύριε Ντεβίγκο. Δεν έχουμε φτάσει ούτε μισή, στα μισά του καταλόγου των ομιλητών. Έχουμε τους ε, σκιώδεις. Ε, σας παρακαλώ όλοι να το έχετε αυτό κατά νου. Ο Ούντο με την ιδιότητα του συντονιστή θα ήθελα να πω στον Πίτερ Σκίνερ τον ε, εισηγητή από την ομάδα μου, τον συγχαίρω για τη δουλειά που έκανε και συγχαίρω και τους λοιπούς εισηγητές φυσικά από τις άλλες ε, ε, ομάδες και θα συμφωνήσω με αυτά που άκουσα. Είναι δυσχερές ε, το έργο, εξαιρετικά περίπλοκο, αλλά έχει κύρια σημασία το όλο εγχείρημα και θεωρώ ότι οι συγητές ήταν εξαιρετικοί. Και έτσι ε, το εγχείρημα θα στεφθεί κατά πάσα πιθανότητα με επιτυχία. Για το θέμα Τέρνερ, δεδομένης της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης που ακόμη βιώνουμε, μπορούμε να πούμε νομίζω ή θα ε, αναθέσουμε ε, μεγαλύτερη αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη ή ευρύτερη αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία, κανένα δίλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχυθεί. Δεύτερον, και όπως είπε εξάλλου και ο Πίτερ Σκίνερ με το σύστημα ελέγχου που προτείνει, η Ευρώπη μπορεί να έχει ισχυρότερα νομοθετήματα μόνο στο μέτρο που κατανοεί την κατάσταση που επικρατεί στις εθνικές αγορές. Πρέπει να κατανοήσουμε τι επιθυμούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να κάνουμε τις απαιτούμενες προσαρμογές, γιατί αλλιώς θα την αποδυναμώσουμε και δεν θα την ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα, ίσως θεωρήσετε ότι υπερβάλλω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη στη συζήτηση που κάνουμε ότι ε, ε, τα κεφάλαια που συγκροτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τελικά, και δεν νομίζω να το θέλει κανείς αυτό, αν τελικά διαμορφωθεί μια κατάσταση όπου οι, οι φορείς εκείνοι, για παράδειγμα, οι τράπεζες ε, και το καθεξής θα πρέπει να διαλύσουν ε, τα ταμεία ασφάλιση τους για να χρηματοδοτήσουν ε, εκείνους οι οποίοι ανέλαβαν λάθος κινδύνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν τους αναγκάσει κάποιες να μειώσουν την ποιότητα των συστημάτων ασφαλεία τους κατά τα συμφερόντων τους θα είχαμε ζημιώσει σημαντικά την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Και είναι σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Σάντσες, ότι θέλουμε την διαφοροποιημένη προσέγγιση των ε, φορέων. Ναι, συμφωνώ, πιο πολύ ενσωμάτωση, όχι πιο πολύ κεντρική διαμόρφωση. Και σε αυτό θα κρυθούν οι εκθέσεις για το κατά πόσο θα τα βγάλουν πέραν με την ισορροπία αυτή για καλύτερη ε, και περισσότερη Ευρώπη αλλά και καλύτερη νομοθεσία όπου θα παραμένουν οι εθνικές αρχές και νομίζω ότι αυτή η διαφοροποίηση, όπως αναφέρατε, βάσει του δυναμικού κινδύνου, θεωρώ ότι είναι ο σωστός δρόμος που θα μας βοηθήσει για την εξέβρεση λύσης. και θα ήθελα να σας καλέσω να συνεχίσετε την δουλειά αυτή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ παραγωγική. Ως σκιώδης εισηγητής για το Συμβούλιο των Κεντρικών Κινδύνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των συστομικών κινδύνων, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Γκουλάρ για την ε, έκθεση του. Νομίζω ότι η κυρία Γκουλάρ ε, κατάφερε να λιάνει, αν θέλετε, κάποια προβλήματα για να καταλήξουμε σε μια καλύτερη νομοθεσία για τους σημαντικούς φορείς από πλευράς ε, χρηστών, αγοραστών, οι γενικοί ενδιαφερόμενοι φορείς που δεν είναι κεντρικές τράπεζες. Θεωρώ ότι είναι σωστή αυτή η προσέγγιση και είναι πολύ σωστό το γεγονό ότι αναφέρεται ότι όλε οι φορεί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να εξεταστούν, όχι να εξαιρεθούν κάποιοι. Αυτό είναι σωστό κατ' ουσίαν. Και επίση συμφωνώ απόλυτα που λέτε ότι χρειαζόμαστε ένα δυναμικό παράγοντα κατά την ανάπτυξη ενό ευρωπαϊκού συστήματο ε, εποπτείας και σε ό,τι αφορά την διαφύλαξη. Και τέλο για το δημοκρατικό έλεγχο, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά αποτελούν προσεγγίσεις που με βρίσκουν ε, σύμφωνο. Παραμένουν κάποια ζητήματα για το ποιος, ε, για παράδειγμα, έχει την ε, εξουσία να προβεί σε προειδοποίηση κινδύνου. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ασάφεια για το ποιος τελικά θα έχει τον τελικό λόγο όταν μιλάμε για εμφάνιση κινδύνου. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε μικρό επίπεδο και μακρό επίπεδο, προκειμένου και σε μικρό επίπεδο να υπάρχει δυνατότητα επισήμανσης κινδύνων στο θέμα της δεσμευτικότητας των αποφάσεων και ποιος είναι υπεύθυνο. Για όλα αυτά θα πρέπει να σας πω ότι ευχαρίστω να συνεργαστούμε μαζί σας, αλλά θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Γιάν Επίνγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω για το την έκθεση της κυρίας Γκουλάρ. Να τη συγχαρώ επίσης για την έκθεσή της. Τη διάβασα με προσοχή. Συμφωνώ με τη δομή την οποία προτείνει. Για το ESRB και για το ESB. Νομίζω ότι πρόκειται για μια προσέγγιση που θα ορίσει καλύτερα τον συστημικό κίνδυνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται συζήτηση για το πώς θα δημορφωθεί η σχετική δομή. Και υπάρχουν ε, ε, αντιθέσεις ε, μεταξύ των δημοκρατών και των συντηρητικών γιατί πλέον έχουν και την πλειοψηφία στη Γερουσία και επιλέγουν άλλη δομή, όχι το Federal Reserve. Οι δομές αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές μεταξύ τους, προκειμένου και εμείς και η ΕΕ να αναπτύξουμε ένα σύστημα το οποίο θα συμβαδίζει με την άλλη πλευρά. Θα ήθελα να σας πω ότι αν ε, διαβρύνουμε το Συμβούλιο σε 67 μέλη ε, θα είναι ήδη υπερβολικό και τους ε, εμπειρογνώμονες στην οι εννέα εμπειρογνώμονες του Συμβουλευτικού α, Επιστημονικού Συμβουλίου που είναι εννέα στον αριθμό και αυτοί είναι πολλοί. Να προσέξουμε. Δεν θα λύσουμε τα προβλήματα επιβάλλοντας γραφειοκρατικό άχθος. σε ένα βιβλίο ενός Αμερικανού πολιτικού αναφέρεται ότι πάρα πολλά ε, αναπτύχθηκαν σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά, ας υποθέσουμε ότι οι τράπεζες ε, έχουν ένα Σαββατοκύριακο στην διάθεσή τους για να επιλύσουν τέτοια προβλήματα. Κανείς δεν πρέπει να πάρει τηλέφωνο, ε, την κυβέρνηση, την διαβουλευτή κτλ. Σε ένα Σαββατοκύριακο πρέπει κανείς να, κληθεί, να πάρει αποφάσεις μετά από πολλά ε, ε, συνελεύσεις. Πρωτού διαλυθεί σε κομμάτια η τράπεζα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια δομή η οποία θα είναι γρήγορη και ευέλικτη. Σε ό,τι αφορά και μεγάλες ε, τράπεζες όπως για παράδειγμα η Deutsche Bank και το καθεξής γιατί θα δημιουργηθεί τεράστια κρατήρα σε περίπτωση έκρηξης τράπεζας τράπεζων τέτοιων. Δεν συμφωνώ με το Advisory Scientific Committee Scientific, επιστημονικό. Τι σημαίνει επιστημονικό σήμερα. Παλιά μαθαίναμε στην οικονομία ότι ήταν ακριβές οι επιστήμες αυτές, ενώ ουσιαστικά αυτό δεν ισχύει τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν βλέπω ποιος είναι επιστημονικός ε, χαρακτήρας. Υπάρχει και η κλιματική επιστήμη, η οποία όπως ξέραμε και αυτή έκανε λάθη. Θα ήμουν προσεκτικός με τη λέξη scientific. Ίσως να σημαίνει κάτι διαφορετικό όμως τα γαλλικά για τις αρμοδιότητες τώρα. Είναι αρκετά οι EPS, οι αρμοδιότητες του ESBRC. D. η και προειδοποίηση. Τίποτα παραπάνω. Μήπως η ESRB θα πρέπει να έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες προκειμένου να μπορεί να αντιδράσει στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχει. Αλλά φυσικά σε την περίπτωση αυτή τη ε, θέμα κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ του ESRB και των τριών ε, αρχών. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχουμε κάνει τη σωστή διάκριση μεταξύ του ESRB και των τριών αρχών αυτών. Ίσως θα πρέπει να μεταφερθούν κάποιες αρμοδιότητες προς το ESRB για να μπορεί να υπάρχει γρήγορη δυνατότητα απόφαση. Αλλά δεν υπάρχει νομική προσωπικότητα του ESRB. Πώς μπορεί να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις. Και τέλος το θέμα του ανοιχτού χαρακτήρα. Αναφέρεται στην έκθεση ότι καμία από τις συστάσεις, ότι το ESRB αποφασίζει αν ε, είναι αξιόπιστες ή όχι. Και παράλληλα αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα θα πρέπει να ενημερώνονται σε περίπτωση που σημειώνεται το τέτοιο περιστατικό. Και σε περίπτωση δηλαδή που η σύσταση είναι απορριτή, εμπιστευτική, κάποια σύσταση για παράδειγμα η οποία θα διαρρεύσει. Όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ σχετικά. Και αυτά θα μπορούσαν φυσικά να διαρρεύσουν και φυσικά αν διαρρεύσουν μια η πληροφορία πάει, καταστράφηκε σε μία μέρα μια τράπεζα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Τι σημαίνει η λέξη απόρριτο, εμπιστευτικό. Τι σημαίνει για μια τράπεζα, για ένα συνταξιδευτικό ταμείο. Γιατί αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο για τα ιδρύματα αυτά, για τα review clause τώρα, για τα ίδρα αναθεώρησης. Αναφέρεται εν μία περίοδος τριών ετών από την Επιτροπή. Εγώ θα προτιμούσα το δύο έτη. Γιατί οικοδομούμε ένα σύστημα το οποίο δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει. Στα αυτοκίνητα, μάλιστα. Έχουμε φτιάξει εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Αλλά το σύστημα αυτό δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Μπορεί και αυτό το σύστημα για την εποπτεία του συστημικού κινδύνου να έχει και αυτό συστημικούς κινδύνους. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα η ρήτρα αναθεώρησης να τεθεί στα δύο χρόνια προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε γρήγορα ενδεχόμενα σφάλματα. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει επαρκής ρύθμιση αγορών και τα συστήματα εποπτείας δεν λειτουργήσαν. Εμείς έχουμε στυλιτεύσει αυτήν την κατάσταση εδώ και καιρό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεύρουμε λύσεις που απαιτούν οι πολίτες. Νομίζω ότι περισσότεροι συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Γι' αυτό τέσσερις πολιτικές ομάδες θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα από τις προτάσεις της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Συμφωνώ με τον Σάντσες Πρεσέδο ότι πρέπει δηλαδή να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Ιδιαίτερα σε σχέση με την αρχή συνταξιοδοτικών αρχών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Όπως είπε ο Σάντσες Πρεζέδο, θα πρέπει να αποφύγουμε μία μελλοντική κρίση. Θα πρέπει να προσδώσουμε μία ευρωπαϊκή διάσταση στο όλο εγχείρημα. Δεν μπορούμε να έχουμε 27 εθνικά εποπτικά συστήματα και ε, δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε ότι είμαστε πολύ μεγάλοι για να αποτύχουμε. Χρειάζεται διασυνοριακή συνεργασία για την αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου. Το παρόν σύστημα εποπτείας δεν μπόρεσε να προλάβει καταστάσεις. Θα πρέπει να μάθουμε πολλά από τα διδάγματα του παρελθόντος και να αναθεωρήσουμε το πλαίσιο ο συντονισμός μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών χρειάζεται. Αλλά αυτό δεν είναι επαρκές. Χρειαζόμαστε μία Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας που να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο και δεσμευτικές αποφάσεις όταν οι εθνικές ε, εποπτικές αρχές δεν συμφωνούν μεταξύ τους και θα πρέπει να είναι άμεσα υπεύθυνη για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αρχών τη στιγμή που πλήττεται η σταθερότητα του συστήματος. Πρόκειται για εποπτεία που θα διασφαλίσουν οι εθνικές αρχές που θα δράσουν κατ' εξουσιοδότηση ακολουθώντας ε, τα, τις υποδείξεις της, Εθνικής Εποπτικής Αρχής, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής, Εποπτικής Αρχής. Επίσης, οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες έναντι καταστάσεων επίγουσας ανάγκες. Επίσης, θα πρέπει να οριστεί ένα ενοποιητικό πλαίσιο μέσα στα πλαίσια ενός νέου, ε, μιας νέας βίβλου κοινών κανόνων που να υποστηρίξει τους καταθέτες στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού εποπτικού συστήματος θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός δράσης σε περίπτωση κρίσης και επίσης ένα ευρωπαϊκό ταμείο όπως πρότεινε και ο συνάδελφος έτσι ώστε οι καταθέτες και οι επενδυτές να μπορούν να διασωθούν και αυτό με βάση τους ίδιους ε, κανόνες του παιχνιδιού για την αποδοτική επίλυση του ζητήματος έναντι ε, παρόμοιων κρίσεων. Βεβαίως υπάρχουν ε, επικρίσεις. Τα μεγάλα προβλήματα όμως χρειάζονται και μεγάλες, μεγάλες εμβέλειες επιλύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να είμαστε φιλόδοξοι στις, ε, στην εποπτεία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα σας πω ποιος περιμένει να μιλήσει. Κλουτ, Πιτέλα. Mrs. Lulling, uh, Mr. Lambert, Mr. Smith and Mr. Tremosa who wants to come back, I imagine, on Omnibus 1. Σε σχέση με το Omnibus 1. Και αυτό είναι το τέλος του καταλόγου των σκιωδών. Ίσως να μην έχουμε χρόνο και να μην μπορέσουν να επανέλθουν οι εισηγητέ. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε στο τέλος. Κλουτ. Ähm, Now. ακούσαμε ήδη και γι' αυτό λοιπόν δεν θα ήθελα να επαναλάβω όσα ακούσαμε. Θα ήθελα να τονίσω κάποιες πτυχές οι οποίες θεωρώ από δικής μας πλευράς ε, ότι είναι σωστές. Καλωσορίζουμε καταρχάς ε, την απάντηση αυτή που προσπαθούμε να δώσουμε στην κρίση σε ό,τι αφορά την εποπτεία των ε, Ιδρυμάτων Αξιολόγησης Πιστοληπτικής ικανότητα θεωρούμε ότι είναι σωστή και ελπίζουμε με τον τρόπο αυτό να περιορίσουμε τον κίνδυνο όντω. Αλλά έχουμε και κάποια σημεία που μας προβληματίζουν. Αναφέρθηκαν ήδη κάποια εξ αυτών. Να τα υποστηρίξω. Σε ό,τι αφορά την κατανομή του προβλήματος των ε, τραπεζικών και λοιπόν ε, τομέων. Πιστεύουμε ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δεν μας φαίνεται πολύ καλή αυτή η διάκριση στο θέμα της διαφάνειας και της αδιαφάνειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά δηλαδή τις διατάξεις για το απόρριτο και την εμπιστευτικότητα θεωρούμε ότι είναι προβληματικές. Θέλουμε ε, ανοιχτό χαρακτήρα για το τι γίνεται και τι προγραμματίζεται. Θεωρούμε ότι είναι βασικό αυτό για να πετύχουμε αυτά που προσπαθούμε να πετύχουμε. Κάτι άλλο, το οποίο δεν το ακούσαμε ιδιαίτερα σαφώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ίσως να υποβάλλεται υπερβολικά σε χρηματοοικονομική εποπτεία. Δεν ξέρω μήπως θα πρέπει να συμπεριληφθούν δηλαδή και άλλες κοινωνικέ ομάδες όπως τα συνδικάτα, όπως ε, οι ενώσεις προστασίας καταναλωτή κτλ. Και επίσης αυτό που μας λείπει είναι ότι θα έπρεπε να έχει το Κοινοβούλιο πιο πολλές αρμοδιότητες. Αυτό θέλουμε να το υποστηρίξουμε. Αυτά λοιπόν, γιατί είναι μακρύς ο κατάλογος των αμελητών και δεν θέλω να, να προβώσω επαναλήψεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιτέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε επτά παρεμβάσεις συναδέλφων εισηγητών που προέρχονται από διαφορετικό γεωγραφικό χώρο και έχουν διαφορετική πολιτική θέση, αλλά υπάρχει ένας κοινό παρονομαστής. Ελπίζω να επιμείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση επειδή στόχος μας ε, είναι η ομοιογένεια και δεν μπορούμε να παλινοδίσουμε θέλουμε να είμαστε συναποφασιστές. Είμαστε ένα κοινοβούλιο που συναποφασίζει και δεν μπορούμε να οπισθοδρομήσουμε έναντι του Συμβουλίου. Έναντι των θέσεων του Κοινοβουλίου, θέσεων που ήταν ιδιαίτερα επιφανειακές. Σε σχέση με τον άνθρωπο Γκίγκολ, το κείμενό του είναι συνεκτικό και συνεπές και πολύ φιλόδοξο διότι θέλει να προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε την κατάσταση. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών των οργανισμών. Είναι ένα θέμα που δεν απασχόλησε κανέναν. Τι θα γίνουν με αυτά, τι θα γίνουν με αυτά τα boards, με τα διοικητικά συμβούλια. Έχουν την ίδια σύνθεση επιτροπών τριτοβαθ, τριτοβαθμίων επιτροπών με εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών. Αυτό αποτελεί αντίφαση με τους αρχικούς στόχους, ε, διότι δεν έχουν επιτύχει αυτές οι επιτροπές, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί υπάρχει μεγάλη αντίσταση από ορισμένες εθνικές εποπτικές αρχές. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει εξισορροπημένη σύνθεση χωρίς να υπάρχουν ε, δεσμεύσεις ή δεσμοί με τις εθνικές αρχές. Αυτή είναι μια υπόδειξη που διαφαίνεται και από την έκθεση de Rozier. Τώρα εντάχει περνάω στα άλλα θέματα. Θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής, θα ήθελα να πω στον εισηγητή, και ως προς τις άλλες οδηγίες, δηλαδή ως προς τα ε, δικαιώματα των μετόχων και την, τον αντικυκλικό χαρακτήρα μέτρων και την ανακύκλωση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι να είναι κοινωνοί αυτής της κατάστασης επίγουσας ανάγκης δυνάμει του άρθρου 12 τροπολογίας 86. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ταμείο χρηματοπιστωτικής προστασίας. Αλλά σε ποιον αποτείνεται, στους καταθέτες ή τους τραπεζίτες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης. Ε, ως προς τη ρήτρα διασφάλισης η τροπολογία 100 υπερβαίνει τον, ε, τον κίνδυνο αυτού του νεφελώματος σε σχέση με το ποιος είναι υπεύθυνος γιατί και πιστεύω ότι η ρήτρα διασφάλισης δεν θα πρέπει να υπάρχει στο κείμενο διότι στην περίπτωση της ΕΣΜΑ ε, δεν υπάρχει καμία επίπτωση επιθεμάτων εθνικής κυριαρχίας. Γι' αυτό θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις να αποκλείονται από τη ρήτρα διασφάλισης. Θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία και στο κεφάλαιο των παραγόγων. Εργαζόμαστε για μία οδηγία που να διέπει αυτή την πτυχή και η ΕΣΜΑ θα πρέπει να εποπτεύει και όχι πλέον οι εθνικές αρχές σε αυτή την πλαισίωση. Ευχαριστούμε. Η Άστριντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, ε, ε, θα ήθελα να μιλήσω για το συστημικό κίνδυνο. Είμαι σκιώδες εισηγήτρια. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Γκολάχ, διότι ε, πήγα στην Επιτροπή Γυναικών για να ψηφίσω επί μία ώρα για την αμφιλεγόμενη έκθεση για την προστασία της ε, μητρότητας και γι' αυτό δεν ήμουν εδώ. Καθησυχάζω. Εδώ όλους τους άντρες περιμένουν παιδί γιατί μπορούν να πάρουν άδεια πατρότητας. Ε, το μόνο που λείπει είναι άδεια συνμητρότητας για τις λεσβίες. Και θα τα έχουμε όλα πια. Ευχαριστώ. Ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ προς την εισηγήτρια. Έχετε όραμα, είναι ποιοτική η έκθεσή σας. Χαίρομαι που τα πάμε τόσο καλά η κυρία Γκουλάχ. Και σε συνεργασία με τους λοιπούς όδης, ελπίζω να καταλήξουμε σε καλή συμβαστική λύση και ελπίζουμε να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Στιμικού Κινδύνου ένα βασικό πυλώνα του μελλοντικού ευρωπαϊκού συστήματος ε, σχετικά με το αν χρειάζεται μια τέτοια αρχή, αν χρειάζεται οργανισμός ε, μα ε, οικονομικής προληπτικής εποπτείας νομίζω ότι έχει λήξει η συζήτηση. Δεν νομίζω κάποιος να αμφισβητεί πλέον την ανάγκη ίδρυσης αυτής της αρχής. Ε, βάσει της έκθεση και της ομάδας Λαροζιέ νομίζω ότι βετεύθη η συνένεση. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο πρέπει να διαμορφωθεί η αρχή, ούτω ώστε να εκπληρώσει τις αποστολέ που θα τις ανατεθούν. Πώς ε, αυτή η Επιτροπή θα λειτουργήσει εύρυθμα σε καθημερινή βάση. Δεν θα ήθελα τώρα να ε, είμαι άκαμπτη γιατί είναι σημαντικό να ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά κάποιων προτάσεων που υποβάλλει η συγγήτρια. Πάντως, ε, γενικά θα έκρινα χρήσιμο πριν μπούμε σε λεπτομέρειες να κάνουμε μία συζήτηση επί της αρχής. Εγώ προτιμώ προς τη σύνθεση της Επιτροπής να προσανατολιστούμε προς ένα περιοριστικότερο σχήμα χωρίς να θέλουμε να τους ικανοποιούμε όλους και τις πεθερές τους όπως λέμε στα γαλλικά ε, πρέπει να μην δημιουργήσουμε ένα γραφειοκρατικό τέρας που θα δυσλειτουργεί. Ε, έχω νομίζω δικαιολογημένους φόβους για αυτό το θέμα και ανησυχίες. Δεν πρέπει ε, να είναι επίσης μονολυθική η Επιτροπή και να αποτελείται από ε, άτομα που όλοι έχουν τις ίδιες ιδέες και τα ίδια πιστεύω. Ε, τέλος, ε, όλοι οι εμπειρογνώμονες ε, του χρηματοπιστωτικού φορέ πρέπει να ακουστούν. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου μόνο μέσα από μια αποτελεσματική λειτουργία θα δίνει χρήσιμες συστάσεις. Αυτή είναι η επιτακτική ανάγκη για μένα και άρα ε, θα πρέπει να είναι άριστη η διαχείρισή της. Τώρα κάτι άλλο για την ΕΚΤΕ και για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών με το, ε, την πρόταση της ομάδας Λεροζιέρ κατευθυνόμαστε προς ε, μία αποκεντρωμένη δομή. Πρόσφατα συγκροτήθηκαν ε, τρεις ε, οργανισμοί ανεξάρτητοι που θα εποπτεύουν τις εθνικές αρχές. Τώρα ως προς την προληπτική εποπτεία βασικό ρόλο θα έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι αιτιολογημένο αυτό δικαίως. Ναι, κατά τη γνώμη μου, η ΕΚΤ. Ας το αναγνωρίσουμε. Ενδυναμώθηκε από την κρίση που μόλις βιώσαμε και στον κύριο Τρίσε επανειλημμένα το έχουμε πει. Δεν είμαι και τόσο πεπισμένη για το διάδοχό του βέβαια. Ε, πάντως πέρασε από το βάπτισμα του πυρός και τα κατάφερε και η ΕΚΤ μπορεί να φέρει σε πέρας και άλλες ε, αποστολές στο μέλλον. Ε, είναι ένα ε, θεσμικό όργανο που καταδεικνύει τον επαγγελματισμό του και νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε σαφώς. Πάντως, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να έχει κέριο και κεντρικό ρόλο ο οποίος ε, αιτιολογείται από το ότι χρειαζόμαστε ένα ε, στοιχείο που οδηγεί στην ολοκλήρωση, σε αντιδιαστολή δηλαδή με τα εθνικά συμφέροντα. Το σύστημα που θέλουμε τώρα να θεσπίσουμε ελπίζω να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών μας. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι η μελλοντική ευρωπαϊκή εποπτεία δεν ε, θα ρυθμίζεται από ένα απλό σύστημα. Χρειαζόμαστε γερά θεμέλια και δεν μπορούμε να ενθαρρύνουμε και στοιχεία. Η ΕΚΤΕΦ έχει ε, βασικό ρόλο να διαδραματίσει, διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο. Η κυρία Γκουλάχ έκανε κάποιες προτάσεις ε, για τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου. Ε, μας μίλησε για την έδρα της Επιτροπής που ενδεχομένως θα είναι στη Φραγκφούρτη. Γιατί όχι. Να το σκεφτούμε. Ε, μπορούμε να κάνουμε και άλλες προτάσεις. Εγώ πάντως ε, προτίθεμαι να το συζητήσω με τους συναδέλφους από την ομάδα μου και με τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές. Λίγη υπομονή ακόμη, ε, Πρόεδρε, για τους υπόλοιπους κανονισμούς σχετικά με την χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπερβεί ε, την παρέμβαση του Συμβουλίου. Το σύστημα που οικοδομούμε αναμφισβήτητα θα μετεξελιχθεί τις, ε, τα επόμενα έτη και σίγουρα που να ακολουθήσουμε την οδό της ε, μεγαλύτερης ολοκλήρωσης και να το λάβουμε αυτό υπόψη όσο εργαζόμαστε στο Κοινοβούλιο γιατί δεν είναι και θέσφατα, όλα, δεν είναι θέσφατες οι προτάσεις που μας έχει δώσει το Συμβούλιο, όλα μπορούν να αλλάξουν. Ευχαριστούμε. Ε, Φιλίπ Λάμπερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία σημεία. Καταρχήν να απαντήσω στη Βίκη για την ανάγκη για τους επόπτες να γνωρίζουν την αγορά πολύ καλά. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να δράσουμε με ταχύτητα. Γνωρίζουμε τις αλλαγές και υπάρχει μια πραγματική ανάγκη, αλλά δεν γνωρίζουμε τις αγορές και τόσο καλά. Εγώ προέρχομαι από μια μικρή χώρα όπου ο καθένας ξέρει το γείτονά του. Και αυτό ισχύει και για το ρυθμιστή που ξέρει τους πάντες σε μια τράπεζα. Και δεν ξέραμε τι θα γίνει, κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει με τη φόρτις γιατί εδώ μιλάμε για συστημικό κίνδυνο, δηλαδή ε, ένα συγκεκριμένο αντίκτυπο και ο ρυθμιστής δεν ήξερε τι συμβαίνει. Ίσως είδε κάτι αλλά δεν ήθελε να το πει γιατί όλοι είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Πρέπει λοιπόν να αποστασιοποιηθούμε διότι εγώ προέρχομαι από μία μεγάλη πολυεθνική και οι επόπτες ήταν πολύ μακριά και όλοι τους φοβόντουσαν. Ναι, πρέπει να φοβόμαστε τις αστυνομικές αρχές, τους επόπτες, γιατί εδώ μιλάμε για μια εποπτική αρχή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοια εγκύτητα με τις εποπτικές αρχές, διότι τότε δεν θα μπορέσουμε να δράσουμε πραγματικά. Νομίζω ότι σε, αυτό το, σε αυτή την περίπτωση το κέντρο βάρους είναι εθνικό και θα πρέπει να υπάρξει μια αποκέντρωση Ε, έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο μέχρι ότου φτάσουμε σε μια ασφαλή απόσταση μεταξύ εποπτικών αρχών και των εποπτευόμενων. Θα ήθελα επίσης να σας μιλήσω για αυτό το θέμα της απαγόρευσης. Το ζήτημα είναι γιατί να περιορίσουμε την για παράδειγμα, α κοιτάξουμε τα χημικά. Απαγορεύουμε προϊόντα. Και γιατί το κάνουμε αυτό. Επειδή δεν ξέρουμε, δεν θέλουμε οι καταναλωτέ να απορροφήσουν και να καταναλώσουν τοξικέ ουσίε. Και τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν τοξικά χρηματοοικονομικά προϊόντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην απαγόρευση, για την απαγόρευση προϊόντων. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι, ξέρετε, χρειαζόμαστε ε, οικονομική δημιουργικότητα, γιατί αυτό βοηθάει την εύρυθμη λειτουργία τη αγορά. Έχω ακούσει αυτό το επιχείρημα εκατοντάδες φορές και θα ήθελα να σας ρωτήσω όλους σας. Έχει λάβει ποτέ κανείς ε, κάποια επιβεβαίωση του ισχυρισμού αυτού. Εγώ ποτέ δεν έχω λάβει κάποιον τέτοια απόδειξη πέρα από αυτή την, ε, τον ισχυρισμό. Πάντα λείπει η δεύτερη και η τρίτη και η τετάρτη και η πέμπτη πρόταση. Αντιθέτως, πλέον έχουμε αποδείξει ότι κάποια προϊόντα αντί να βοηθούν την εύρεθμη λειτουργία της αγοράς, καταστρέφουν τη λειτουργία αυτή. Αν θέλουμε λοιπόν να βασίσονται οι πολιτικές μας σε γεγονότα και συγκεκριμένα, συγκεκριμένα στοιχεία, θα πρέπει να τα εξετάσουμε τα στοιχεία αυτά. Και παρεπιπτόντως, οι τράπεζες παραδέχονται ότι ούτε και αυτές καταλάβραν, τι πουλούσαν. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρξει σωστή εποπτεία, πώς θα καταλάβουν οι, υποπτή, οι αρχές τα προϊόντα που δεν καταλαβαίνουν καν αυτοί που τα πουλάνε. Αν θέλουμε να λειτουργήσει η εποπτεία, θα πρέπει να εξετάσουμε την λύση απαγόρευσης προϊόντων. Και τέλος, κάτι σε σχέση με την διαδικασία. Και εδώ, Βίκυ, μίλησες και εσύ σε ό,τι αφορά την νομική βιωσιμότητα των θεμάτων. Και θα ήθελα να μιλήσω για την τροπολογία 138 του πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες, όπου υπήρξε ευρεία συμφωνία, ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο. Αλλά γεγονός είναι ότι η τροπολογία 138 που υποστηρίχθηκε από το 88% του Κοινοβουλίου ήταν ουσιαστικά χωρίς σωστή νομική βάση. Δεν θέλω λοιπόν να προκύψει μια σειρά εκθέσεων οι οποίες σε τελική ανάλυση να μην αντέξουν μετά τη νομική εξέταση, γιατί στην περίπτωση αυτή θα γελιοποιηθεί το Κοινοβούλιο στα μάτια του Συμβουλίου, γιατί επειδή θα ακολουθήσει που θα ακολουθήσει η σύγκρουση με το Συμβούλιο, θα ήθελα να διασφαλίσω και ας χρησιμοποιήσουμε την νομική μας υπηρεσία και οτιδήποτε χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ό,τι θα γράψουμε στις εκθέσεις αυτές θα στέκει και θα αντέξει στην κριτική του Συμβουλίου. Αυτό πρέπει να το κάνουμε για να μην γελιοποιηθούμε στις επόμενες φάσεις της διαδικασίας. Ευχαριστώ, κύριε Σόλου Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντα υποστήριξα το 1 3 και στο τέλος φτάσαμε σε ένα πολύ καλό συμβιβασμό. Και στις ε, ευρωεκλογές έπρεπε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, ορισμένες προτάσεις μας πάντα θα θεωρούνται οι μη παράνομες από μερικούς. Περίεργη παρατήρηση αυτή. Πρόκειται για μία τεράστια πρόκληση. Από τότε που μπήκα στο Κοινοβούλιο το 1999, ε, μπορώ να πω ότι επιτελέσατε μία εξαιρετική εργασία και μερικοί συνάδελφοι το σκέφτηκαν αυτό νωρίτερα. Η Έκε Βάντεμπεργκ το 99-2000 άρχισε με κάτι τέτοιο και μετά είχαμε ένα φιλελεύθερο συνάδελφο κατά την τελευταία θητεία. Θα πρέπει να τους θυμίσουμε διότι προείδαν την κατάσταση. Είμαι υπέρ της διαφάνειας βεβαίως, αλλά νομίζω θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν λέω ότι απορρίπτω αυτά που προτείνεται, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα καταρτήσουμε, το καταρτήσουμε λίγο καλύτερα αυτό το πλαίσιο, διότι η διαφάνεια μπορεί να είναι αντιπαραγωγική. Μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες και απορρίτου χαρακτήρα. Κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί επιζήμιο για επιχειρήσεις και για χώρες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ορισμένες ε, επιχειρήσεις. Και αυτό ε, λέχθη από τον κύριο Έπινγκ. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς τις διαρροές αυτών των πληροφοριών. Θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλιά σας επ' αυτού. Γιατί μπορεί να σταθεί πραγματικά επιζήμιο. Υπάρχουν ε, μικρές χώρες και δεν υπάρχει τόσο υψηλό συστημικός κίνδυνος σε αυτές τις χώρες. Ίσως μπορεί να υπάρχει ειδική στοχοθέτηση και αυτό ήταν το παράδειγμα σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσφατα. Το Ταμείο Σταθερότητας τώρα, ως προς αυτό, θα πρέπει να υπάρχει μια μελέτη αντικτύπου και δεν θα ήταν συνετό να απορρίψουμε το όλο πλαίσιο και να πούμε ότι δεν μας ε, ταιριάζει. Και το ως προς τον κύριο Λάμπερτ που είπε ότι θα πρέπει να απαγορέψουμε προϊόντα. Ναι, υπάρχουν επιχειρήματα. Α, έφυγε και ο κύριο Λάμπερτ. Σω καλά έκανε, πολύ καλά έκανε. Α, είναι παρόν. Αχ, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, σα κατέκρινε. Άλλαξε θέση, αλλάξατε θέση. Θα έπρεπε να είσαστε ιδιαίτερα ευτυχεί ω φιλελεύθερο. Όποιο είναι κοντά στου φιλελεύθερου θα πρέπει ε, να θεωρήσει τον εαυτό του ευτυχή. Λοιπόν, αν δεν κατανοείτε τα προϊόντα, πώς μπορείτε να τα απαγορεύσετε, αν δεν τα κατανοείτε. Θα πρέπει να υπάρχει ευέλικτη προσέγγιση διαφορετικά. Θα πρέπει να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Αρχή Απαγορεύσεων που κάθε εβδομάδα θα πρέπει να απαγορεύσει κάτι. Έτσι δεν είναι. Κάτι λέει ο άλλος βουλευτής εκτός μικροφώνου. Προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτά που είπατε και τις συνέπειές τους. Το ρίστο το ψηφίσατε εσείς, αντιτείνει ο άλλο βουλευτής. Τώρα μιλάμε για απαγόρευση προϊόντων στον χρηματοοικονομικό τομέα. Κύριε Λάμπερτ, μιλήσατε. Μην παρεμβαίνετε σαν να είμαστε σε νηπιαγωγείο. Δεν λέω ότι αντιτάσσομαι σε όλες τις ρυθμίσεις. Αλλά ακούσετε με, υπάρχουν ε, ε, προβλήματα και αν πληγεί ένα τομέα, θα προχωρήσουμε στον άλλον. Θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, εξεταστικοί ως προς κάθε προϊόν. Κάθε δηλαδή καταναλωτής θα μπορεί να λέει, ε, να έρχεται κάθε εβδομάδα και να σας λέει «Α, απαγορεύσε αυτό το προϊόν». Εγώ πρέπει να μπορώ να βασίζομαι σε αυτά τα προϊόντα. Θέλω να είμαι ένας υπεύθυνο καταναλωτής. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε κανονισμούς. Υπάρχει μία ε, χρηματοοικονομική εκπαίδευση και στη χώρα μου. Αλλά όταν μιλάτε για απαγόρευση προϊόντων, δεν ξέρετε ποια προϊόντα απαγορεύεται, δεν τα κατανοείτε. Και αυτό είναι περίπλοκο. Ακούσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία σφραγίδα ποιότητας. Δηλαδή μία Ευρωπαϊκή Αρχή να ορίζει την ποιότητα. Δεν νομίζω ότι είναι συνετή η ιδέα αυτή, γιατί θα ήταν πολύ περίπλοκο. Δεν λέω όμως ότι φταίτε για όλα γιατί είμαι φιλελεύθερος. Γιατί θεωρώ ότι όλοι ή σχεδόν όλοι έχουν ε, ψίχουλα σοφίας. Πολύ μεγάλη πρόκληση λοιπόν και νομίζω ότι ήταν ε, εξαιρετική η εργασία σας και ελπίζω ε, εμείς τα πίσω έδρανα που δεν είμαστε ούτε καν σκιώδεις να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο ο Σε κάτι, σε κάτι λέει η πρόεδρος. Μακάρι να ήξερα σε τι. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό θα μιλήσω. Ο Σκιώδης για την ε, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια όχι μόνο για την εργασία της, αλλά για τον ε, προευρωπαϊστικό χαρακτήρα της έκθεσής της. Θα πρέπει να εξεύρουμε μηχανισμούς εποπτείας αγοράς, γιατί καταγγέλουμε την κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια ως Κοινοβούλιο. Η πρώτη ανάγνωση είναι καλή. Προσπαθούμε να ε, βελτιώσουμε την ε, χρηματοπιστωτική αρχή. Προσπαθούμε να έχουμε μία ευρωπαϊκή αρχή η οποία να στυλιτεύει τις εθνικές εποπτικές αρχές όταν σφάλουν. Αυτή τη φιλοδοξία τη συμμερίζομαι και αυτό αφορά και περισσότερους της ομάδας μου. Σε σχέση με τα διασυνοριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο εισηγητής θεωρεί θα πρέπει να δώσει περισσότερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή και προτείνει περισσότερη εσωτερική αγορά και λιγότερο προστατευτισμό. Αυτή είναι και ο συστή ο οδός, λαμβάνοντας υπόψη την εποπτεία μεγάλων χρηματοπιστωτικών αρχών. Στην ομάδα μου λαμβάνουμε υπόψη και την ευαισθητοποίηση του εισηγητή σε σχέση με την χρηματοδότηση των ΜΜΕ όπου ε, συμμετέχει και το Συμβούλιο Εποπτικής, ε, Εποπτικών Αρχών. Και θεωρούμε ότι όταν σφάλουν οι τράπεζες θα πρέπει να κατακρίνονται το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβάλλει μια πρόταση έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή αρχή με σαφείς αρμοδιότητες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αρχικές προτάσεις de la Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον Oui, Madame merci. Euh, θα ήθελα να δώσω ορισμένε διευκρινήσει στον κύριο Λαμπέρα, αλλά βλέπω ότι μιλάει, μιλάει. Α, θα με ακούσει από ό,τι φαίνεται. Ω προ την απαγόρευση των προϊόντων. Καθόλου κακή ιδέα. Κάθε αυτή. Μπορώ να σας πω όμως, επειδή βρισκόμουν σε ένα πιστοτικό ίδρυμα, ότι οι γαλλικές αρχές ε, δεν δέχτηκαν κάτι τέτοιο γιατί αποτελεί μεγάλη διοικητική ευθύνη. Άρα η ρυθμιστική αρχή δεν μπορεί εκ των προτέρων να εξετάσει τα προϊόντα αν υποθέσουμε ότι τα ε, κατανοεί για να ξέρει κατά πόσο είναι τοξικά ή όχι. Επίσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι η χρηματοπιστωτική δημιουργία δεν προσθέτει τίποτα. Τώρα το ζήτημα είναι κατά πόσο τη συγχαίουμε με κάτι άλλο. Νομίζω όμως ότι πολλές χρηματοδοτήσεις δεν θα γίνονταν αν δεν υπήρχε χρηματοπιστωτική δημιουργικότητα. Πρέπει όμως να χαλιναγωγείτε. Είπατε ότι θα πρέπει νομικά να είμαστε σταθεροί και στεναροί. Σας λέω όχι η ρύθμιση ως προς τα ιδρύματα πιστοληπτικής ικανότητας, ε, ως προς την προηγούμενη έκθεση είχαμε 600 τροπολογίες και στην Επιτροπή συμφωνήσαμε μαζί με όλους τους συναδέλφους για μία διάταξη που να λέει ότι η εποπτεία των οργανισμών πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Αλλά νομικά δεν ευσταθεί αυτό. Άλλος, κάποιος άλλος όμως είπε ότι είναι πολιτικά αναγκαία. Ε, όμως νομικά δεν ήταν εφικτό. Όταν βρεθήκαμε στον τριμερή διάλογο με την ε, Κομισιόν και την Τσεχική Προεδρία τότε, μου είπαν ότι νομικά δεν γίνεται. Εγώ τους είπα όμως ότι κατά μία μεταβατική φάση, ας κάνουμε αυτό που λέτε, αλλά θα πρέπει να δεσμευτείτε να αλλάξετε τους κανόνες για να καταστεί εφικτό και σήμερα στο κείμενο για την αρχιτεκτονική εποπτείας, εκεί η μόνη ευρωπαϊκή εποπτεία αφορά τους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας. Δεν θα είναι πολύ υψηλή αυτή η εποπτεία, αλλά ψηφίσαμε κάτι το οποίο νομικά δεν ήταν δυνατό και μας επέτρεψε στις ε, διαπραγματεύσεις να υποστηρίξουμε την Επιτροπή. Δεν χρειάζεται να είμαστε ε, στην ουσία ε, να εμένουμε σε ορισμένα ζητήματα εκεί που δεν έχουμε λόγο. Έχουμε 10 λεπτά μόνο και πολλούς ε, εισηγητές. Δεν ξέρω κατά πώς θα τα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Θα ακολουθήσω την άλλη σειρά, την αντίστροφη σειρά Αν, αν το δεν θέλει το λόγο εντάξει. Η Σιλβή. Πολύ σύντομα. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που σχολίασαν. Πολύ καλές ιδέες παρουσίασαν. Ως προς το δικό μου κείμενο υπάρχουν ε, πολλά σημεία που χρήζουν εργασίας το θέμα της διαφάνειας και του βαθμού διαφάνειας σε σχέση με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα αποτελεί μία λεπτή ισορροπία. Μπορώ να το δεχτώ αυτό, υπάρχουν όμως κοινοβούλια που ασχολούνται με ζητήματα εμπιστευτικού χαρακτήρα και στον τομέα της άμυνας. Θα πρέπει λοιπόν, αν και δεν έχουμε όλα τα μέσα να διατηρήσουμε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιτελεστεί πρόοδος. Ένα άλλο στοιχείο, όπως είπε και η κυρία Λούλινγκ που έφυγε, είναι πώς μπορούμε να δούμε την σύσταση, τη σύνθεση των οργάνων, την τήρηση αρμοδιοτήτων, κανένα πρόβλημα και εκεί. Τέλος, όταν μίλησα για ένα ε, συμβουλευτικό, για ένα συμβούλιο, Επιστημονικό Συμβούλιο, ίσως θα πρέπει να έχουμε κάποιον που να είναι μαθηματικός, ε, υψηλής εμβέλειας μεταξύ των συμβούλων, έτσι ώστε η Sharon Bowles να μπορέσει να θριαμβεύσει. Ίσως χρειαζόμαστε και ανθρωπολόγους και κοινωνιολόγους. Αυτό το πλαίσιο είναι πολύ κλειστό όλα αυτά ήταν, δεν ήταν παρά προτάσεις. Θα ήθελα να πω στους αλλούς συναδέλφους ότι συμφωνώ με το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ίσως θα πρέπει να μας απασχόλησει περισσότερο για να συμφωνήσουμε με το ESRB. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε ένα ανοιχτό διάλογο. Πίτερ. Πίτερ Σκίνερ, ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ ο κ. Ζάλμπερ. Αλλά πρέπει να πω ότι ήταν ενδιαφέρον το ότι προσπάθησε να αποτυπώσει αυτά που συνέβησαν στο τραπεζικό κλάδο, στον ε, κλάδο τον ασφαλιστικό. Ο Χωσέν Μανουέλ είπε ότι ήθελε να κοιτάξει την ε, σωστή προσέγγιση για το 2,5% του ΑΕΠ αλλά στις ε, ασφαλίσεις και στις συνταξιοδοτήσεις τι θα σήμαινε αυτό για το ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Νομίζω ότι μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα για τις ε, συντάξεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2011. Μπορείτε να, μπορεί να μου πείτε, μπορεί να μου απαντήσει κανείς. Ίσως να βγούμε έξω και να αρχίσουμε να ζητάμε χρήματα. Από αύριο. Μπορούμε να ζητήσουμε στις αρχές αυτές να πληρώσουν για κάθε ευρωπαϊκό σφάλμε. Δύσκολο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ανέφικτο. Δεν πιστεύω ότι είναι εφικτό, αλλά ας ε, θέσουμε ε, τη φιλοδοξία αυτή Θεωρείτε, κυρία Γκάουσες, ότι πρόκειται να πληρώσει το Παρίσι για λάθος των Βρυξελών, να του ζητήσουν να πληρώσουν και για τα σφάλματα του Ηνωμένου Βασιλείου και θα δείξουν την ίδια διορία. Οι πρακτικές πλευρές λοιπόν θα πρέπει να λεφθούν υπόψη για τη δημιουργία ενό ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, για το FSA ε, μιλάμε για προσωπικό 3.000 ατόμων. Υπάρχει πλήρες ε, καταρτισμένο, πλήρως καταρτισμένο προσωπικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είμαι κατά της αρχής. Απλά θεωρώ ότι στην πράξη, για να εφαρμοστεί που από Ιανουαρίου 2011, ε, η οδηγία για το CR θα τεθούν σε εφαρμογή χωρίς ε, άλλα νομοθετήματα. Ε, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Ας μην κοροδευόμαστε. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν τι θα κάνουμε σε ό,τι αφορά τη φάση της εφαρμογής της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν και άλλοι τρόποι από το να επιτρέψουμε το Συμβούλιο να κάνει τι θέλει, κοιτώντα τις κοινέ επιτροπές για το πώς μπορούμε να δεσμεύσουμε τους ε, υπαλλήλους να αντιδράσουν μαζί με όλα τα σώματα για να δημιουργήσουμε την ισορροπία που επιθυμούμε. Αν απλά μιλήσουμε για μεγάλες φιλοδοξίες, για ανέφικτα σχέδια για τον συνταξιδοτικό και ασφαλιστικό κλάδο, δεν θα καταφέρουμε αυτό που πετύχουμε. Να είναι πρακτικές οι φιλοδοξίες μας, να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Να έχουμε υπόψη τις πρακτικές πτυχές του Solvency 2 και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε για να συνεργαστούν οι ρυθμιστικές αρχές ως ενιαίο σύνολο. Δεν θέλουμε αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τις φιλοδοξίες μας. Γιατί αν θέλουμε να το παρεκβάλλουμε αυτό και σε άλλους κλάδους, μπορεί να με λειτουργήσει στους άλλους κλάδους. Ο Σβέν, λέει η Πρόεδρος. Ναι. Κάτι έμαθα και σήμερα. Dass die, ε, dass mein Vorurteil ότι η προκατάληψη που είχα για τους συντηρητικούς και για τους χριστιανοδημοκράτες ε, ότι αγαπούν την τάξη δεν αληθεύει. Ότι μπορεί κανείς να υποβάλει προτάσεις που δεν είναι καν νόμιμες. Και όλα αυτά από νομικούς. Με δισκετάζει ιδιαίτερα το γεγονό αυτό. Και χαίρομαι που αυτό ανησυχεί και άλλα άτομα. Μοναδικό αυτό στην Επιτροπή μας, να πω. Όχι, όχι. Ε, κάνω δωρεά σε ένα ίδρυμα για την υποστήριξη κοινωνικών ε, κινημάτων. Να σχολιάσω για κάποια στοιχεία μόνο. Καταρχάς, το θέμα της επικουρικότητας. Νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα ότι η αρχή αυτή της χριστιανικής ηθικής πάντα α, τη χάνει κατάχρησης για να πετύχουμε τους πολιτικούς μας στόχους. Σωστή η αρχή της επικουρικότητας, αλλά δεν θεωρώ ότι σημαίνει ότι όλα θα πρέπει να περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο. Όχι. Να είναι τόσο τοπικά όσο χρειάζεται. Και αν κάτι έχει αποδειχτεί από την κρίση αυτή είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στις διασυνεριακά εντρήματα. Αν υπάρχει δίκτυο εθνικών εποπτικών αρχών, υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ε, αποτελεσματική τους δράση σε εθνικό επίπεδο. Άρα, όπου υπάρχει ισχυρή παράδοση τοπικής ε, εποπτικής αρχής και τοπικών εποπτικών δερμάτων δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ευρωπαϊκή εποπτεία. Χρειαζόμαστε έναν κοινό κώδικα, αλλά όχι να εξευρωπαίσουμε, αν θέλετε, τη διαδικασία αυτή. Όταν όμως μιλάμε για, τα μεγάλα, για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς, η δομή φαίνεται ότι δεν επαρκεί. Λέγοντας λοιπόν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2011 και με τα επιχειρήματα αυτά και πώς θα βρούμε το, το προσωπικό, ε, ποτέ δεν θα είχαμε καταλήξει στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα που έχουμε σήμερα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το επιχείρημα. Είναι σημαντικό λοιπόν η μεγάλη διασυνοριακοί θεσμοί και οι επόπτες να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε ρυθμίσει πρακτικά τι σημαίνει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ότι χρειάζεται για παράδειγμα ε, χιλιάδες ε, άτομα προσωπικό. Θεωρώ ότι τα ευρήματα απεστροπτικής ικανότητα και κάποιοι άλλοι θεσμοί θα το κρίσουν αυτό. Τέλο, για την απαγόρευση των προϊόντων, δεν πρότεινα να απαγορέψουμε ό,τι δεν αρέσει στου πράσινου. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Οι οικονομικές αγορές θα πρέπει να είναι καινοτομικές και πρέπει να παραμείνουν καινοτομικές. Δεν λέω ότι θα πρέπει να απαγορευτούν όλα τα προϊόντα, επειδή δεν το καταλαβαίνω εγώ ή ο Φίλιπ. Όχι, δεν πρότεινα κάτι τέτοιο. Αυτό που πρότεινα είναι το εξή, ότι υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία αποδείχθηκαν επιζήμια και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, το δικαίωμα εκ μέρους της ΕΣΜΑ να τα απαγορεύσει, αν χρειαστεί. Και θα έλεγα ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με πολύ επιφυλακτικό τρόπο μιλώντας για παράδειγμα για τις ακάλυπτες πωλήσει, ότι είναι ε, επικίνδυνες. Αν απαγορευτεί στη Γερμανία, αυτό θα ασκήσει και στις άλλες αγορές. Μάλλον, αν επιτραπούν αυτές οι πωλήσει στη Γερμανία, αυτό θα ασκήσει και σε άλλες αγορές για να τις επιτρέψουν εκ νέου. Αν λοιπόν θέλουμε υπό συγκεκριμένου όρους να απαγορεύσουμε κάποια προϊόντα τα οποία έχουν αποδειχθεί επιζήμια σε όλες τις αγορές, όχι σε μία μόνο, θα πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η Πρόεδρος μας είπε, η Πρόεδρος λέει ότι οι διερμηνείς συμφώνησαν να δώσουν πέντε λεπτά παραπάνω. Να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον κύριο Μαγκάλο. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ η Βίκη Φόρτ σε σχέση με, για να μιλήσουμε για την μεθοδολογία εργασίας, διότι θα θέλαμε να υπάρξει εσωτερική συνοχή μεταξύ εκθέσεων που άπτονται διαφορετικών ε, ζητημάτων σε σχέση με το τι λένε οι διάφορες ε, πολιτικές ομάδες. Τη στιγμή λοιπόν που έχουμε ένα κοινό λιμπρέτο θα πρέπει να δούμε από κοινού ε, μία σειρά τροπολογιών. Δεύτερον, ως προς το θέμα μίας ισχυρής ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής και αυτής της εξισορρόπησης με το θέμα της λογοδοσίας, accountability. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε έναν μικρό κατάλογο. Είναι σαν να έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό beauty contest. Δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί η συζήτηση που είχαμε ως προς το νομισματικό διάλογο με τον πρόεδρο της ΕΚΤ. για ότι η ΕΚΤ και η Αρχή Ανάληψης Συστημικού Κινδύνου θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα με ε, μία πρόβλεψη 15 ημερών, δηλαδή ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές, ποιοι επόπτες δεν ακολούθησαν το σχέδιο, ποιοι έπρεπε να επιπληχθούν και ούτω καθεξής. Όλα αυτά υπάρχουν στην έκθεση. Ο Ραμόν Τρεμόσα που ήταν γενναιόδωρος, ιδιαίτερα γενναιόδωρος, μίλησε για τη σύνθεση. Βεβαίως, η έκθεση για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ασχολήθηκε με τις τράπεζες και όχι με όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εδώ σκέφτομαι ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, διότι η μεγάλη επιχειρήση μπορεί να έχει ροή κεφαλαίων πιο εύκολα. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι η πρόληψη και η ενημέρωση των εποπτικών αρχών, δηλαδή ποιο είναι το κόστος αυτής της πίστοσης για τις ΜΜΕ, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ροή. Και εμείς είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό. Λέμε λοιπόν ότι σε αυτήν την ομάδα ενδιαφερομένων θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση, πολυπληθής εκπροσώπηση των ΜΜΕ και να συμμετέχουν και στο Συμβούλιο Εποπτικής Αρχής έτσι ώστε η χρηματοπιστωτική οικονομία να υπηρετεί την πραγματική οικονομία. Με ρώτησαν μερικοί για το τι θα γίνει ως προς τις τραπεζικές αρχές. Δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ. Μιλώ για το Turner Review που μίλησε για την Ισλανδική κρίση. Έχει σημασία η επιχείρηση έδρα σε σχέση με τη θηγατρική γιατί πολλές φορές οι επόπτες που βρίσκονται στις θηγατρικές δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτό το κίνδυνο και καταβάλουν το κόστος. Και η καγκελάριος, καγκελάριος μας είπε ότι δεν μπορούν οι τράπεζες που μας οδήγησαν στο γκρεμό να συνεργαστούν με βρετανικές τράπεζες για να αντιμετωπίσουν χρηματοπιστωτικές κρίσεις όπως η ελληνική. Πολλές φορές ελέγχθη ότι φταίει η νεοσυντηρητική σκέψη ως προς την εποπτεία. Επίσης, μιλήσαμε για ένα πλαίσιο κυρώσεων και θα ήταν κρίμα οι αγορές που μας ε, οδήγησαν στον ε, γκρεμό να, είναι αυτές, να μην είναι αυτές που θα καταβάλουν το κόστος, αλλά να το, καταλάβουν, να το καταβάλουν άλλες. Το Συμβούλιο πόρο απέχει από τις θέσεις ε, του Κοινοβουλίου. γιατί ε, θυμάμαι την περίπτωση ενός σταυρομάχου που βρισκόταν στο Μπορντό και ο οποίος ε, είπε ότι θα έπρεπε να βρίσκουμε η Σεβίλη. Η Σεβίλη είναι μακριά και του ελέγχθη όχι. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Δεν είναι μακριά το Μπορντό από τη Σεβίλη, αλλά η Σεβίλη από τον Μπορντό. Αυτό αφορά την απόδοση ευθυνών. Και έχει σημασία η τροχοπέδη που υπάρχει για να φτάσουμε στο, στην τσέπη του φορολογούμενου. Στην ΟΝΕ είδαμε πολλά ερωτήματα. Στην έκθεση Βέρνερ το είδαμε αυτό. Ε, γιατί ο κύριος Σάμουελσον στη Μαδρίτη είπε ότι να μπει η Ισπανία στην ΟΝΕ σημαίνει να πάει κανείς και να κοιμηθεί με έναν ε, ε, γορίλα. Είναι τόσο δηλαδή παράδοξο. Αυτό είχε πει τότε ο κύριος Σάμουελσον. Δηλαδή ε, αυτά τα παράδοξα γίνονται. Ναι εντάξει, εντάξει, θα συγκρατηθώ. Θα συγκρατηθώ, αν και δεν τα καταφέρνω πάντα. Δυσκολεύεται και τους διερμηνείς, εκτός από όλους τους άλλους λέει η πρόεδρος. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε με το χρονοδιάγραμμα. Θα το διανύμουμε, αλλά θα έχουμε το ίδιο, το, το ίδιο χρονοδιάγραμμα αυτό που έχετε ήδη. Αργότερα αυτή η εβδομάδα θα μιλήσουμε για την κατάσταση της Ελλάδας και τις προειδοποιήσεις του Συμβουλίου. Η προειδοποίηση εδόθη δυνάμει του άρθρου 121 τη συνθήκη της Λισαβόνας και γι' αυτό θα ασκήσουμε, θα ε, ακολουθήσουμε αυτό το δικαίωμα. Η παράγραφος 5 του 121 θα ζητήσει από το Συμβούλιο να έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου για δημόσια συστάσεις. Θα στείλω αυτή την επιστολή αύριο.